και την ομιμότητα των πληρωμών εκτός από τις... Ε, ήταν λοιπόν η μόνη υπηρεσία, η ΕΑΣΟ, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη από το ηλεκτρικό συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν να ανασταλούν οι πληρωμές. Το δικαστήριο εξέδωσε μία ε, απόφαση σύμφωνα με την οποία ε, αναφέρθηκε σε μη συμμόρφωση της ΕΑΣΟ με τις διαδικασίες ε, προσλήψεων μεταξύ άλλων. Το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΑΣΟ για το οικονομικό έτος 2017. Αυτό σημαίνει ε, δηλαδή ότι αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΑΣΟ για το 2017. Αποφάσισαν λοιπόν να ε, να παγώσουν λογαριασμοί από τότε και στο εξή. Εμείς προτείνουμε ω ε, Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού κατόπιν εξέτασης των ακολούθων διαπιστώσαμε μέσα στα ευρήματα, παρατυπίες σε σχέση με τη ε, διαδικασία προσλήψεων, κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων, κατάχρηση εξουσίας, παραβιάσεις των, ε, του κανονισμού προσωπικών δεδομένων, ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό και περιπτώσεις παρενόχλησης. Επίσης, η συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση δείχνει μία ανεπαρκή ικανότητα εσωτερικού ελέγχου στην ΕΑΣΟ. Η κυρία Γκρεγόρη, η οποία είναι τώρα εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού, μας είπε πως δεν υπήρχε εσωτερικό σύστημα ελέγχου της υπηρεσίας το 2017. Επίσης, υπήρξε ένα συνδυασμό σφαλμάτων που ε, οδήγησε σε μια απώλεια της ε, τάξης του 10 περίπου της 100 του συνολικού προϋπολογισμού του οργανισμού. Με την ιδιότητα του εισηγητή για την απαλλαγή της ΕΑΣΟ πρέπει να τονίσω ότι ο προϋπολογισμός για το 2017 εκτελέστηκε υπό την εποπτεία της προηγούμενης διοίκησης της ΕΑΣΟ και αυτή η έκθεση που εξετάζουμε σήμερα αφορά τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017. Μετά, υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ ενδιαφέρον για όλους στην Ευρώπη. Η νέα διοίκηση της ΕΑΣΟ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διορθώσει τα λάθη της προηγούμενης διοίκησης. Αυτό δεν ήταν θαύμα, αλλά ήταν αντικείμενο και αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Κανείς δεν περίμενε να γίνουν θαύματα σε μία νύχτα, όμως έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Πριν από δύο χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς ε, θα μπορούσαν να διορθωθούν τα πράγματα. Και να είστε σίγουροι, επειδή παρακολουθώ πολύ στενά την ε, περίπτωση αυτή, το 2018 που ξεκίνησαν ε, κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες. Επιθυμούμε η παρούσα διοίκηση να συνεχίσει τις ε, προσπάθειές της και να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Θα υπάρχει και παρακολούθηση της ε, έκθεσης και εμείς στηρίζουμε απόλυτα το σχέδιο δράσης το οποίο μας έχουν δώσει από τη δίκηση της ΕΑΣΟ. Μάλιστα τον Ιούνιο μας ε, έστειλαν και την πέμπτη επικαιροποιημένη εκδοχή του σχεδίου δράσης. Είμαστε σίγουροι ότι η ΆΣΟ θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και θα συμμορφωθεί με τις ε, συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Επίσης, καλωσορίζουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο προσλήψεων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Σίγουρα υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα να διανύσει η Άσο, όμως είμαστε σίγουροι πως όλα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να συνοψίσω, η Άσο με τη σημερινή της μορφή δεν έχει καμία σχέση με την Άσο πριν από δύο χρόνια. Όμως, σήμερα έχουμε κληθεί να ασχοληθούμε με την απαλλαγή του 2017 και όχι ε, του 2019. Γι' αυτό να πω ότι πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας στα σοβαρά. Εάν χορηγήσουμε απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2017 στην ΕΑΣΟ, για μένα θα πετάξουμε στα σκουπίδια την όλη έννοια της άσκησης απαλλαγής. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και θα έστελνε λάθος μήνυμα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Λάθος μήνυμα από τον, ε, στον απλό πολίτη, ε, στον ε, διευθυντή, σε άτομα που χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια μέχρι τους κοινοτικούς μηχανισμούς, τους ενωσιακούς μηχανισμούς. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη, διαφορετικά θα καταρρεύσει. Αυτό είναι και το νόημα τούτης της απαλλαγής. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία για την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από εκείνα τα προβληματικά χρόνια μέχρι τώρα και για την απαλλαγή στην στη διοίκηση εκείνη του 2017. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να δεχτούμε, ε, να χορηγήσουμε μια τέτοια απαλλαγή χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρη η διαδικασία απαλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πέτρη για τη σκληρή δουλειά σου. Τώρα, θα περάσω από τον εισηγητή στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Είναι μία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που έχουμε να εξετάσουμε. Ε, θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στην Ελέωρα Βόλτας. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για το σχέδιο έκθεσης για ένα ζήτημα που είναι πολύ πιο πολύπλοκο από μια απλή απαλλαγή. Είναι περίπλοκη έκθεση γιατί επισημαίνει τις ε, δυσκολίες του παρελθόντος, αναγνωρίζει όμως ταυτόχρονα και τα θετικά ε, μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έκτοτε και όπως λέει βέβαια και η έκθεση πρόκειται για την απαλλαγή του έτους 2017. Αυτό πρέπει να το έχουμε συνεχώς υπόψη. Ταυτόχρονα για μένα τίθεται το εξής ερώτημα το προηγούμενο κοινοβούλιο πήρε την απόφαση αναβολής της απαλλαγής ε, παρότι τότε ε, ήδη ήταν ε, παρελθόν το 17. Γιατί λοιπόν πριν τις θερινές διακοπές δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί απόφαση. Φαντάζομαι η απάντηση είναι ότι έκτοτε λήφθησαν νέε πληροφορίε υπό μορφή του εγγράφου που έστειλε η Άσο με τα μέτρα που έχει λάβει, αλλά Υπήρξε στο μεταξύ και η εκτίμηση της Όλαφ, στην οποία έχουμε πρόσβαση. Εγώ προσωπικά θέλω να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε χρόνο να μελετήσουμε τα δύο νέα αυτά έγγραφα και μετά να λάβουμε απόφαση. Εγώ προσωπικά θέλω να έχω λάβει γνώση των δύο εγγράφων και να μπορούμε ε, περιστατωμένα να πάρουμε μια απόφαση. Ε, πραγματικά είμαι διχασμένη αυτή τη στιγμή. Βλέπω και αντιλαμβάνομαι την πολυπλοκότητα Τη υπόθεση αυτή. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει σοβαρή δουλειά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ξακολουθήσω να μελετώ αυτό το θέμα και με χαρά να συνεργαστούμε και με εσά και με τους υπόλοιπου συναδέλφου. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ραμόνα, εσείς τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με τα λόγια της αντέλφου. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω. Πολύ περιεκτική πλήρηση δουλειά που έχετε κάνει και θα μας βοηθήσει πολύ. Και πρέπει να συνεχίσουμε στο πνεύμα που αναφέρατε εσείς προηγουμένως και συγητά. Ακριβώς ε, σε χάρη των προσπαθειών που καταβάλουν όλα τα θεσμικά οργανά για τη διαφάνεια, για τη χρηστή διακυβέρνηση, για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων ή οποιασδήποτε παρατυπίας ή κατάχρησης ε, των κονδυλίων που ουσιαστικά είναι χρήματα των φορολογουμένων. Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο η μελέτη του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, ε, που εκτούμε ιδιαίτερα από την διοίκηση, για να μπορέσει να εφαρμοστεί με σωστό ενδεδειγμένο τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος, χρειάζεται έλεγχος, παρακολούθηση και εφόσον πλέον διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα γίνονται με τον σωστό τρόπο, θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε μια διαφορετική πιο ευνοϊκή απόφαση. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και τίποτε περισσότερο. σας ευχαριστώ πολύ. Κράμουν. Ευρύτερα, δηλαδή υπό το πρίσμα της πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται ένας οργανισμός που να λειτουργεί σωστά. Μας έκανε μια πολύ αναλυτική και πλήρη παρουσίαση και επεξήγηση κατάστασης η νέα διοίκηση. Προς το παρόν δυσκολεύονται να προσλάβουν, να προσελκύσουν επαρκές προσωπικό, προσωπικό που χρειάζεται. Υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό δίλημα. Διότι εάν δεν χορηγήσουμε απαλλαγή για το 2017 στην ΝΑΖΟ, τα πράγματα θα καταστούν ακόμη πιο δύσκολα. Να είναι δηλαδή καθαρή εντός εισαγωγικών υπηρεσία, άσπηλη στην εικόνα της και να πέσουν στην παγίδα υποψήφια που θα θελήσουν να γίνουν ε, μέλη του προσωπικού ε, αυτής του οργανισμού που βαρύνεται με το παρελθόν αυτό, τα πολλά σκάνδαλα και τις παρατυπίες. Είναι, αν θέλετε, βρώμικο το παρελθόν του οργανισμού. Πρέπει να καθαρίσει. Με το σχέδιο δράσης λύνονται τα περισσότερα προβλήματα. Εκκρεμούν 13 ακόμη, αλλά αν κατάλαβα καλά, εργάζεται από αυτόν η υπηρεσία, άρα και αυτά θα λυθούν. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Άρα, θα πρέπει να δούμε σαν μεμονωμένη και μοναδική περίπτωση την κατάσταση του έτους 2017, που φυσικά και θα πρέπει να μελετηθεί, να διερευνηθεί, να την παρακολουθήσουμε. Όμως, εγώ θα συνιστούσα αντίθετα από τους προηγουμένους ε, να εγκρίνουμε το δεύτερο σχέδιο έκθεσης Δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε για τη μη χορήγηση. Έχετε ζητήσει και εσείς το λόγο, ε, κύριε Κούρς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε και νομίζω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ακριβώς ε, τι λέει και ο κανονισμός του Κοινοβουλίου που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να χορηγήσει απαλλαγή και έχουμε και το 261 άρθρο στο πρώτο εδάφιο που λέει ότι η απόφαση περί απαλλαγής έχει να κάνει ε, τον υπολογισμό όλων των εσόδων, εξόδων και την καθάριση όλων αυτών. Δηλαδή μιλάμε για οικονομικά ζητήματα. Αυτά που μας δημιουργούν προβλήματα δεν έχουν να κάνουν τόσο ε, με, ή τόσο αποκλειστικά μόνο με τα οικονομικά. Αν κατάλαβα καλά, ε, από οικονομικής πλευράς είναι εντάξει τα πράγματα. Τέλο πάντων έχουν όλα διευθετηθεί σε ό,τι αφορά δηλαδή τους λογαριασμούς και επομένως ε, αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Εκεί που υπήρξαν προβλήματα ήταν ε, οι ιστορίες αυτές παρενόχλησης ε, και ασημνής ανάρμοστης της κτλ. κτλ. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτό, τέλος πάντων υπάρχει ένα αποτέλεσμα και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απαλλαγής άμα αφήσουμε να φέρει αυτό το βάρος, ε, τα πράγματα θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται. Άμα κουβαλάνε αυτό το στίγμα και άμα τους πούμε δεν ήσασταν καλοί, δεν τα κάνατε καλά, δεν έχετε διορθώσει την κατάσταση, δεν μπορούμε να σας δώσουμε απαλλαγή. Εγώ νομίζω αυτό θα ήταν ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό θα συνιστούσα πραγματικά να χορηγήσουμε απαλλαγή το 2017 και όλα τα άλλα θέματα που αναφέρονται και στην έκθεση και που έχουμε διαβάσει τα πορίσματα και τα οποία ε, βλέπουμε και στις εκθέσεις άλλων οργανισμών, να τα μελετήσουμε ώστε να δοθεί και σε αυτά ένα αίσιο πέρας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. θα πρέπει ίσω να συζητήσουν ξανά οι συγκητές με του και συγκητές ό,τι αφορά ε, την απαλλαγή, γιατί αφορά το 2017 και πρέπει να δούμε τι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και βέβαια σίγουρα δεν μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση ή κάτι τέτοιο, αλλά και το κατά πόσο κάποιο υποχρεώθηκε να κάνει κάτι δεν υποχρεώθηκε έχει να κάνει, έχει παίζει κάποιο ρόλο για την οικονομική εκαθάριση, για ε, το κλείσμα των λογαριασμών. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να γίνει μια συζήτηση. Να παρακαλέσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ΠΕΑΤΕ ε, να πει ορισμένα πράγματα, αλλά έχω και εγώ μια ερώτηση. Ε, νομίζω και άλλοι ίσως διερωτήθηκαν τι γίνεται με αυτό τον κατάλογο ε, με τις ε, παραλήψεις και τα λάθη που ε, θα μπορούσε να γίνει στη Γερμανία δίκη για όλα αυτά. Εδώ δεν υπήρξε κάποια δίωξη και πραγματικά εμένα αυτό με ανησυχεί γιατί εγώ βλέπω ε, να υπάρχουν ποινικέ ε, επιπτώσεις. Ε, δηλαδή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο οικονομικά ζητήματα. Για μένα έχει και ποινικέ διακλαδώσεις και συνέπειες. Υπάρχει αυτός ο κατάλογος που εμένα με παραπέμπει και στο ποινικό κώδικα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση. δεν είναι τόσο ελάσσονα αυτά τα αδικήματα και αυτές οι συμπεριφορές. Και αυτό που είπε η Βιόλα των Κράμων, ίσως η Κομισιόν δεν μπορούσε να απαντήσει, αυτή η μεταπίδηση υπαλλήλων από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Υπήρξαν τέτοιου είδους ε, καταγγελίες. Και ο πρόεδρος στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Home ήταν σε μια άλλη ε, θέση. Πώς έγινε αυτή η μεταπίδηση και πώς προτάθηκε για τη θέση του Διευθυντή από την Κομισιόν. Συμπληρώνω αυτή την ερώτηση και την ε, στρέφω στην Επιτροπή ουσιαστικά για αυτήν απευθύνεται, νομίζω και όχι στην κυρία Γκριγκόρη που δεν μπορεί να απαντήσει. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν. Και τώρα έχετε, κύριε και Μπεάτε, έχετε μία πολύ απλή ε, δουλειά να κάνετε, να απαντήσετε τα πολύπλοκα αυτά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνατε τη δυνατότητα να εκφραστώ. Ονομάζομαι Μπέατε Κμίντερ, υπεύθυνη οικονομικής διαχείριση από την ε, Γενική Διεύθυνση Home. Ασχολούμαι λοιπόν με εσωτερικά ζητήματα. Τώρα, δεν μπορώ ακόμα να απαντήσω στην ερώτησή σας για τον λόγο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εξέτασης της περίπτωσης αυτής. Σε ό,τι αφορά την ε, πειθαρχική διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο του, ε, της ΕΑΣΟ είναι αρμόδιο για να επιβάλλει ε, τις ε, κυρώσεις στον πρώην εκτελεστικό διευθυντή. Τώρα, η σχέση διακυβέρνηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των οργανισμών αυτών είναι. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κυρίω συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έχουμε προτείνει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν κατάλογο. Βέβαια, αυτό έγινε προτού αναλάβω καθήκοντα, οπότε δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά για το περιεχόμενο. Ε, το μόνο που ξέρω είναι ότι την εποχή εκείνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε άλλον ε, υποψήφιο ε, στον οποίο είχε δείξει προτίμηση για τη θέση αυτή. Όμω, ο τότε εκτελεστικό διευθύντη ανέλαβε καθήκοντα κατόπιν ε, πλειοψηφία του Συμβουλίου. Τώρα, η διαδικασία, ε, η πειθαρχική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει και σε συνέπειες. Μπορεί να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις ή και άλλες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα και δεν μπορώ βεβαίως να απαντήσω στην ε, ερώτησή σας. Όμως ε, να σας ευχαριστήσω ξανά για αυτήν την πολύ ισορροπημένη γραμμοδότηση σχετικά με την απαλλαγή για το 2017. Πιστεύω ότι αυτό δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι το έργο της χορήγησης απαλλαγής και σίγουρα πρέπει να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενότατη επαφή με την ΕΑΣΟ για να καταρτήσουν ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα συνοδεύσει. Έχουμε βιντεοδιασκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουμε μάθει πάρα πολλά από την περίπτωση ΕΑΣΟ οι συνάδελφοί μου από τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνοι για άλλους οργανισμούς έχουν αντλήσει διδάγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε το μέλλον να αποτραπεί ε, η επανάληψη μιας ε, τέτοιας ε, περίπτωσης. Πρέπει βέβαια να αναλυφθούν ευθύνε και αυτό να ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον Πέτρη Σαβάρμα όχι έχει το ρόλο του εισηγητή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως επαναλαμβάνομαι, το έχω ξαναπεί. Βασικά το έχω πει δύο φορές, γιατί την πρώτη φορά το είπα και κλεισμένον των θυρών. Αλλά θα το ξαναπώ. Για τρίτη φορά λοιπόν σήμερα. Σημείωσα με προσωπικό τα όσα είπε η Λάρα Βόλτερς. Έχει δίκιο. Όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το ζήτημα αυτό δεν είναι εύκολο, είναι κάθε άλλο από εύκολο. Όμως, σε τελική ανάλυση νομίζω πως ε, θα τελειώσω με αυτά που είπα και πριν. Αυτό που κάνουμε στην Επιτροπή με την άσκηση της απαλλαγής, με αυτές τις εκθέσεις, είναι ένα καθήκον που υπάρχει παντού, υπάρχει στις συνθήκες. Έχουμε την ευθύνη να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος και να χορηγήσουμε απαλλαγή στην περίπτωση αυτή ε, στον εκτελεστικό διευθυντή που έφταιγε για όλη αυτή την κατάσταση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, ε, εγώ το βλέπω κάπως απλά. αυτό, αυτή είναι η δουλειά μας. Αν δεν κάνουμε τη δουλειά, τη δουλειά μας, τότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Τότε θα ζοριστούμε. Και να το θυμάστε, του χρόνου, του παραχρόνου σε μερικές δεκαετίες, ε, δεν θα, θα, θα ξαναρθούμε σε αυτό το θέμα, θα το εξετάσουμε ξανά. Διότι έχουμε την ε, περίπτωση ενός ανθρώπου που παραλίγο να καταστρέψει έναν ολόκληρο οργανισμό και αν το κοιτάξουν οι μελλοντικέ γενιές, τι θα κάνουν, πώς θα το δουν. Αν μετά από 20-30 χρόνια ψάξουμε και να τρέξουμε σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα βρει κανείς τίποτα. Έχει κοντέψει να διαλυθεί ο οργανισμός και δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Μόνο αν ψάξει θα δει ότι κάτι είχε συμβεί. Εγώ δεν, δεν, μπορώ να το δω έτσι όμως το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ε, συναδέλφους που έθεσαν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην κυρία Γκρεγόρη. Ε, όσον οι ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν ακόμα, θα παρακαλέσω να μου τις στείλετε γραπτός, έτσι ώστε να τις διαβάσω στην ε, κυρία Γκρεγόρη. Γνωρίζω πως το ζήτημα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πειθαρχημένη στάση που κρατήσατε. Να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Σεπτεμβρίου. 25-26 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε μάλλον την, στη, δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρεγόρη, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Πραγματικά η Επιτροπή μας αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Γι' αυτό λοιπόν και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια διότι σας χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε γενικά άτομα σαν και εσάς στην ΕΑΣΟ. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εξέταση του δεύτερου σχεδίου έκθεσης. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Απαλλαγή Γενικός Περιπολογισμός της Ένωσης. Η συγκήτρια είναι η κυρία Γκαρθία Μουνιός και της δίνω Στο στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, σύμφωνα με το 319 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η υπεύθυνη αρχή ε, για να εγκρίνει ή να απορρίψει τη διαχείριση της Κομισιόν κατά την εκτέλεση του προπολογισμού. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να επιβεβαιώσει ότι ο προπολογισμό διατέθηκε νόμιμα και ε, νομότυπα με μια ορθή οικονομική διαχείριση. Πρόκειται για μια πολύ βασική αρμοδιότητα τη Κομισιόν προ όφελο των, των όλων των πολιτών τη Ευρώπη και φορολογουμένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία σε δημοκρατικό επίπεδο και το σύνολο του, του προπολογισμού τη Ένωση. Η συνθήκη αναφέρεται στην έγκριση τη διαχείριση τη Κομισιόν για λόγους διαφάνεια και, και δημοκρατικής εποπτείας εγκρίνει και τη διαχείριση ε, ξεχωριστά ε, και για τις άλλες υπηρεσίες ε, της ε, Ένωσης. Εξετάζει λοιπόν τα έγγραφα το Κοινοβούλιο, εξετάζει τις απαντήσεις των ερωτηματολόγια που εστάλησαν, ακούει και τους γενικούς γραμματείς των θεσμικών οργάνων που έρχονται στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Πρόκειται λοιπόν για μια πρακτική η οποία είναι θεσμοθετημένη, το δέχονται όλα τα θεσμικά όργανα, εκτός από το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, από το 2009 το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να εγκρίνει τη διαχείριση του Συμβουλίου λόγω της έλλειψης συνεργασίας από την πλευρά του Συμβουλίου. Στην διαδικασία για το κλείσιμο των λογαριασμών του 2017, που είναι αυτό που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, για άλλη μια φορά το Συμβούλιο δεν μας διαβίβασε τα στοιχεία που του ζητήσαμε έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να εγκρίνει ή όχι τη διαχείριση του Συμβουλίου. Ούτε ήταν παρόν στην ακρόαση με του Γενικού Γραμματεί που οργάνωσε αυτή η Επιτροπή. Έτσι λοιπόν στι 26 Μαρτίου το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ε, ανέβαλε την έγκριση των ε, λογαριασμών του Συμβουλίου στον Οκτώβριο για να του δώσει την ευκαιρία να διορθώσει ε, το λάθος του. Δεν έκανε όμως τίποτα το Συμβούλιο δυστυχώς έως τότε και ω σήμερα δεν έχουμε λάβει ακόμα τίποτα από το Συμβούλιο. Για άλλη μια φορά λοιπόν αυτή η Επιτροπή, εφόσον δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ε, θα απορρίψει τη διαχείριση του Συμβουλίου για το 2017. Η συνθήκη σε ό,τι αφορά ε, της, ε, το Συμβούλιο και τη διαχείρισή του υπάρχει, το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σύστασης. Το Συμβούλιο ε, βεβαίως βασίζεται σε μια συμφωνία κυρίων του 1970 όταν αποφάσισαν ε, ότι θα εγκρίνουν ε, τα δύο αυτά θεσμικά όργανα τους λογαριασμούς το ένα του άλλου αμοιβαία χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί όμως με τέτοια συμφωνία κυρίων να εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. Πρέπει να αντιδράσει το Συμβούλιο, να καταλάβει το δημοκρατικό λόγο, ρόλο που παίζει το Κοινοβούλιο στην περίπτωση αυτή, να αποδεκτεί τον δημοκρατικό έλεγχο των λογαριασμών του όπως συνέβη για, το, για τα άλλα θεσμικά όργανα. Όλα, αυτά τα χρόνια έγιναν πολλές απόπειρε και από τα δύο θεσμικά όργανα έτσι ώστε να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας. Δυστυχώς ε, δεν οδήγησε αυτό σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσει που διακόπησαν ουσιαστικά πριν από ένα χρόνο διαπραγματεύσει κατά τη διάρκεια των οποίων η Επιτροπή μας πρέπει να παίξει έναν θεμελιώδη ρόλο και που πρέπει να βασιστούν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένα κοινό έδαφος που να σέβεται τις αρμοδιότητες και των δύο θεσμικών οργάνων ε, προ όφελο των πολιτών της Ευρώπης. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω το Συμβούλιο να είναι διατεθειμένο να φτάσει σε μια συμφωνία για να συνεργαστούμε το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, στην έκθεσή μου αναφέρομαι επίσης σε κάποιες από τις πτυχές των λογαριασμών του Συμβουλίου, το οποίο υπογραμμίσαμε και στην έκθεση του Μαρτίου. Υπάρχει ανησυχία, διότι είναι ε, αυξημένα τα κονδύλια τα οποία έχουν μεταφερθεί από το 2018. Θα πρέπει ε, να υπάρξει διαχωρισμό ε, σε δύο δημοσιονομικέ γραμμέ του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία και θεσμικά όργανα και βεβαίω να διευκολύνουμε και τον έλεγχο των δαπανών. Και τέλο, υπάρχει ανάγκη για μια πιο ευέλικτη διαδικασία για να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το μητρό ε, διαφάνειας. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε ένα ζήτημα το οποίο έχει βγει και στον τύπο στην Ευρώπη και που απασχολεί τους συμπολίτε μας. Πρέπει να μας απασχολεί λοιπόν όλους, ιδιαίτερα σε ένα πλαίσιο όπου τα θεσμικά όργανα, οι θεσμοί ευρωπαϊκοί χρειάζονται την εμπιστοσύνη, χρειάζονται την ενίσχυση της εμπιστοσύνη των πολιτών και αναφέρομαι στο θέμα των ιδιωτικών sponsorship. Πολλά κράτη-μέλη το κάνουν αυτό όταν αναλαμβάνουν την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό για κάποια χρόνια ήταν η εξαίρεση. Πλέον όμως είναι ο κανόνας. Το Συμβούλιο πολλές φορές μας έχει απαντήσει ότι ο προπολογισμό της Προεδρίας είναι ευθύνη του κράτους μέλους που έχει αναλάβει την Προεδρία. Ακόμα και σε ό,τι αφορά την, το, τους ιδιωτικούς ε, σπόνσορες. Παρότι αυτό δεν είναι παράνομο, θα, θε, θα συμφωνείτε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ε, αξιοπιστίας, διαφάνειας, εμπιστοσύνης απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην δώσουμε την εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, οι πολίτες δεν μπορούν να διαχωρίσουν τόσο εύκολα θεσμικά όργανα μεταξύ του Συμβουλίου, παραδείγματος χάρη και τη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, είναι ένα θέμα λοιπόν που αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα το ίδιο το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα απλά σήμερα να σας, να σας διαβιβάσω την ανησυχία μου έτσι ώστε να γίνει μια συζήτηση, η οποία είναι δημόσια πλέον βέβαια, μιας και θεωρώ ότι από πολιτικής πλευράς είναι καλό να το αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση. Από την πλευρά μου, εγώ προβλέπω να προσθέσω μια τροπολογία εντός της προθεσμίας που προβλέπετε και βεβαίως ε, ε, σας ενθαρρύνω, ενθαρρύνω τα μέλη της Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους, να αποφύγουμε πάνω απ' όλα να χρησιμοποιηθεί αυτό το θέμα από τους λαϊκιστές για να επιτεθούν την αξιοπιστία της ε, Ένωσης. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην πρώτη σκιώδη συγγήτρια, την συνάδελφο Βίντσικ. Χαίρομαι που είναι και ο κύριος Γιάκοψα ε, ο κύριος Γιάκοψ από το Συμβούλιο εδώ. Για να τα σημειώσει όλα και να τα μεταφέρει. Και Ρία, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρθία Μουνιώθα, την εισηγήτρια για την εργασία της ως εισηγήτρια από πλευράς του ΕΛΚΑ. Στηρίζω πλήρως ε, την έκθεση και ελπίζω και εγώ να βρεθεί σύντομα λύση για τι διαφορές αυτέ που έχουμε με το Συμβούλιο και να τηρηθεί αυτή η συμφωνία ε, κυρίων ε, που δεν είναι πλέον αναλογική. Και σίγουρα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοχή και εμπιστοσύνη από του Ευρωπαίου πολίτε προ τα θεσμικά όργανα. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε και την επιστολή της κύρια Κολμάιερ που έστειλε στι 26 Ιουλίου στο Συμβούλιο και στην επιστολή αυτή για μια ακόμη φορά η κυρία Χολμάγερ. μιλά για το non-payer του Ιουλίου του 2018, αυτό το ανεπίσημο έγγραφο και ζητά εκεί ε, να τοποθετηθεί το συμβουλευτό. Θέλουμε να περιληφθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σαστέλ. Είστε ο τρίτος ε, στη σειρά σκιώδης Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και εγώ την κυρία Γκαρθία Μουνιώθ για το σχέδιο έκθεσης. Όπως είναι προφανές, από την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να αλλάξει στάση ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε ως, ε, όπως προηγουμένως ε, στη θέση μας και να μην χορηγήσουμε απαλλαγή στο Γενικό Γραμματεία του Συμβουλίου για την εκτέλεση του προπολογισμού για το οικονομικό του 2017. Και νομίζω ότι αυτό σίγουρα είναι επιζήμιο ε, στην ε, στάση του Συμβουλίου, ότι αρνείται το διάλογο δηλαδή συστηματικά. Ελπίζω ε, να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ και κάποια χρόνια, το 2009 το περιμένουμε βέβαια και δεν το βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε να καταλάβει το Συμβούλιο ότι έχει ε, νόημα να σεβαστεί την πρακτική που σέβονται όλα τα άλλα θεσμικά όργανα. Και έτσι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι εμπιστεύονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι μακρύς ο πράγματι διότι την άρνησή μα, όπω είπε και η συγγήτρια, την αιτιολογούμε βάσει του ότι δεν μα έδωσε απαντήσει στο Συμβούλιο στι γραπτέ απαντήσει. Ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου δεν παρίστατο στην ακρόαση του Νοεμβρίου 18, στο πλαίσιο τη διαδικασία ετήσια απαλλαγή. Το Συμβούλιο δεν απάντησε στι παρατηρήσει που είχε διατυπώσει στο ψήφισμα τη 26η Μαρτίου 2019 για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο και το Μάρτιο του 19 το Κοινοβούλιο ήδη είχε αρνηθεί την απαλλαγή στο Γενικό πράγματα του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017. Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ θερμά είναι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με το Συμβούλιο για να εξελιχθεί κατάσταση, αλλά δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να αλλάξουμε εμείς θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους πρασίνους είναι ο συνάδελφος Πεξάης. Um, uh, uh, in what uh, my... Να συνεχίσω κι εγώ στην ίδια γραμμή με τους προλαλήσαντες. Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε τη θέση μας όταν ε, η θέση του Συμβουλίου παραμένει η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ. Ωραία. Ωραία, και εγώ λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Αστέλ, ελπίζω να βγούμε γρήγορα από αυτό το αδιέξοδο και να καταφέρουμε, να προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να συνεννοηθούμε, διότι ε, πράγματι πρόκειται για προϋπολογισμό του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ας ε, προσπαθήσουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε εδώ την κατάσταση και ίσως ε, να φερθούμε ως ενήλικες και να δείξουμε την ε, κατανόηση και τη συμπεριφορά που πρέπει. Ελπίζω λοιπόν μαζί με την ε, εισηγήτρια και με όλους εσάς, τους σκιώδεις εισηγητές, να το καταφέρουμε, να το προσπαθήσουμε, έστω ε, άλλη μία φορά. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας στηρίξω ως πρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Κλούκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η τρίτη συνεδρίαση στην οποία παραβρίσκομαι και διαπιστώνω με τρόμο ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αναρωτιέμαι αν αυτή η κατάσταση τραβάει τώρα εννέα χρόνια και υπάρχει αυτός ο αρνητισμός, τι μπορούμε να κάνουμε ε, πέρα από το να συζητάμε. Αυτό δηλαδή θέλω να ρωτήσω. Έχει το Κοινοβούλιο κάποια δυνατότητα να κόψει κονδύλια από το Συμβούλιο? Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αν το μόνο που έχουμε είναι η συζήτηση, τότε πάντα σε τείχο θα πέφτουμε. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Ναι, πρέπει να δείξουμε κατανόηση και πρέπει να ρωτήσουμε όμως και τα ουσιώδη. Δηλαδή, τι νόημα έχει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγή όταν δεν έχουμε πρακτικά κανένα δικαίωμα άσκηση πίεση. Αυτό σκέφτομαι τις τελευταίες ε, ημέρες έτσι, που έχω έρθει σε αυτές τις συνεδριώσεις. Ε, νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ότι πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται. Όταν οι συζητήσει δεν οδηγούν πουθενά, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει, πρέπει να γίνει και το μπαμ. Να το μάθει, να το μάθει ο κόσμος. Έστω και αν αυτό ακούγεται έτσι πολεμοχαρές, αν ακούγεται λαϊκιστικό, ε, κάποια στιγμή πρέπει να το, πει και, να το πούμε κιόλα έτσι. Ωραία. Η κυρία Φων Η ε, κυρία Φων είχε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, δημιουργική πρόταση. Όμως, όπως και να έχει, αναφέρθηκε από την Αγγέλικα αυτή η συμφωνία κυρίων. Δεν πρόκειται για συμφωνία. Ε, το μόνο που έχουμε συμφωνήσει είναι να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός, όλα τα υπόλοιπα δεν υφίσταται. Πάντα υπήρχε λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων να μην ε, μπλέκουμε στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και αντίστοιχα το Συμβούλιο σέβεται τις ε, προτάσεις του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό μπορείτε να τα βρείτε όλα, είναι, υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Αυτό ε, είναι το ζητούμενο. Και σίγουρα το Συμβούλιο έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες και ανάγκες για προσωπικό, διότι μην ξεχνάτε το Συμβούλιο αποτελείται από 28 κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν οφείλει και να προστατεύει το Κοινοβούλιο από πολιτικές πιέσεις, αλλά εμείς πρέπει να προστατεύουμε και τα συμφέροντά μας. Εμείς δεν έχουμε ούτε Συμβούλια Υπουργών από πίσω, ούτε 28 ε, κρατημέλη, ένα όργανο είμαστε. Βέβαια, όλα τα πάντα, όλα τα στοιχεία είναι ε, δημόσια. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Και νομίζω πως αυτή η έκφραση συμφωνία κυρίων είναι λανθασμένη, δεν είναι η σωστή διότι δεν υπάρχει τίποτα συμφωνημένο έτσι και κλεισμένο των θυρών, ούτε παρασκηνιακά, όλα είναι διαθέσιμα, ανοιχτά. Και να δούμε ποια είναι η επικοινωνία την οποία έχει το Συμβούλιο μαζί μας σε θέματα απαλλαγής, σε θέματα προϋπολογισμού. διότι ακούγεται συχνά ότι το Συμβούλιο μας ε, κρατά διάφορα κρυφά, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Εγώ πάντως σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να επικοινωνήσω με το Συμβούλιο έτσι για να προχωρήσει το θέμα όπως ε, γίνεται και με τους άλλους ε, οργανισμούς, όπως γίνεται και με την Επιτροπή των Περιφερειών και τα ε, άλλα θεσμικά, με τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ζητούν απαλλαγή από εμάς. Ελπίζω λοιπόν πολύ σύντομα να σταματήσει λοιπόν αυτό το πρόβλημα, να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε μια λύση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω εδώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητέ. Ας ξαναπροσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι, θα γίνει. Ωραία, 10 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Έγκριση, ε, ψηφίζουμε στην Επιτροπή 23-24 Σεπτεμβρίου και δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Τώρα περνάμε στον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 όλα τα τμήματα και περνάμε στην εισηγήτρια Κορίνα Κρέτσουτη, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που θα παρουσιάσω σήμερα το έργο μας γύρω από την έκθεση αυτή για το οικονομικό έτος 2020. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ο προπολογισμός αυτός για το επόμενο δημοσιονομικό έτος είναι το, τελευταίο, το τελευταίος στο παρόν πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα προπολογισμό που θα είναι και ένας προϋπολογισμός συνέχειας αλλά και μετάβασης. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που σας υποβάλλω αφορά όλα τα τμήματα του προπολογισμού, όλα τα κεφάλαια. Θα αναφερθώ μόνο σε κάποια σημεία τα οποία έχουμε ενσωματώσει, κάποιες προτάσεις που προέρχονται από εσά και από τη γραμματεία, όπως η οικονομική διαχείριση και τις σχετικές δηλώσεις προγραμμάτων για τις δαπάνες και ε, τα έσοδα, ε, μετανάστευση, οικονομικά εργαλεία και βεβαίως το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, Ευρωπαϊκός Αγγελία, Έχετε λάβει το σχέδιο γνωμοδότηση από τη γραμματεία. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη ό,τι αφορά τις αλλαγές που προτείνουμε σήμερα. Ε, για την οικονομική διαχείριση θέλω να υπενθυμίσω ότι ο 247, το άρθρο 247 του κανονισμού αναφέρεται στην υποχρέωση τη Κομισιόν να ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο και, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο μάλλον μια έκθεση ε, λογοδοσίας. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτή η έκθεση να αναφέρεται στις δεσμεύσεις και στο ποιος είναι ο αντίκτυπός τους, ε, τι γίνεται με τις καθυστερήσεις στα πλαίσια του πολιτισμού του δημοσιονομικού πλαισίου. Σε σχέση με την προγραμματική δήλωση για τις επιχειρησιακές δαπάνες, ε, καλωσορίζουμε τη δήλωση αυτή για το έτος 2020 μας δίνει πληροφορίες ε, για το, κάθε, για το καθένα από τα προγράμματα ε, δαπανών. Θα πρέπει όμως ε, η Επιτροπή Προπολογισμού από κοινού με άλλες επιτροπές αυτού του, του, του Κοινοβουλίου να προωθήσουν μια κουλτούρα που να βασίζεται στο αποτέλεσμα να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των χρημάτων και να ζητήσουμε περισσότερα μέτρα για καλύτερη απορροφητικότητα και αποδοτικότητα. Το λέω αυτό διότι είμαστε πλέον στο 2020, έξι χρόνια έκλεισαν από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε αργή εφαρμογή. Χθε ο Γενικός Διευθυντής στην DG Regio παρουσίασε αυτή την αργή εφαρμογή των προγραμμάτων λιγότερο από 30% του προπολογισμού του 2014-2020 έχει δαπανηθεί και ανησυχώ. Ανησυχώ διότι υπάρχει πειρασμός από τα κράτη-μέλη ε, να υπάρξουν προγράμματα, ή project, ε, μόνο και μόνο για να λάβει χώρα απορρόφηση. Δεν σας κρύβω ότι σε, πήγα σε πολλές χώρες και είδα ότι είναι μια πρακτική αυτή τα τελευταία χρόνια, τις τελευταία, της πραγματικής περίοδου, να γίνονται, να σχεδιάζονται προγράμματα μόνο και μόνο για την απορρόφηση, χωρίς να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς δείκτες για το πώς δαπανώνται αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Ε, σε ό,τι αφορά την, ε, τις εκθέσεις απόδοσης και το streamlining πρέπει να λάβει η χώρα. Έχετε δει τους διάφορους δείκτες ε, για την κάθε έκθεση απόδοσης. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους δείκτες εκείνους που μετρούν καλύτερα την απόδοση ε, του κοινωνικού προπολογισμού και επίσης ε, ε να μάθουμε κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί αυτοί οι δείκτες για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την απόδοση. Υπάρχει ένα στόχος να έχουμε μια πλήρη και δίκαιη εικόνα για το τι επετεύχθη θα πρέπει λοιπόν οι εκθέσει αυτέ για την απόδοση όταν χρειάζεται να οδηγούν σε διορθωτικά μέτρα όταν δεν πληρώνονται οι στόχοι. Επίση πρέπει να παρουσιάζουμε σαφώ πληροφορίε για, τα, για τι προκλήσει που μένουν να απαντηθούν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα τώρα εξακολουθώ να ζητάω από την Κομισιόν να υπάρχει ακρίβεια σε ό,τι αφορά τις ε, προβλέψεις για τις δαπάνες, ε, να μάθουμε από το παρελθόν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, ε, διότι πολύ συχνά τελικά υπάρχει συμφόρηση ό,τι αφορά τις μένει, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, γιατί τη μετανάστευση δεν πήρα το λόγο νωρίτερα όταν συζητήσαμε την υπηρεσία, την ΕΑΣΟ, το θέμα της ΕΑΣΟ. Αυτό που προτείνουμε είναι να έχουμε ένα ξεχωριστό δημοσιονομικό, δημοσιονομική γραμμή για, τον στόχο, για τους στόχους του προγράμματος Δάφνη, να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ζητούμε αυξημένους πόρους για αυτή τη δημοσιονομική γραμμή. Εγώ προσωπικά θα υποστηρίξω αυτή την τροπολογία, ελπίζω να με ακολουθήσετε, διότι αυτή η ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή σε αυτό το προπολογισμό αφορά μόνο μετανάστες κοριτσιά, μικρά κορίτσια, ανήλικους που έρχονται από τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να κλείνουμε όμως τα μάτια ε, σε αυτό που συμβαίνει και στα δικά μας κράτη-μέλη, στην Ήπειρό μας, στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα είχαμε μια τραγωδία πολλά νεαρά κορίτσια που δολοφονήθηκαν. Από ό,τι φαίνεται υπήρχε ένα δίκτυο που είχε ε, διασυνδέσεις και σε άλλες χώρες. Ε, θέλουμε λοιπόν υποστήριξη για να υπάρχει μια τροπολογία για να προστατεύουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια όχι μόνο για τους μετανάστες ε, αλλά να καταπολεμήσουμε την εμπορία ανθρώπων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρότασή μου για τα οικονομικά μέσα τώρα. Βεβαίω οι συζητήσει συνεχίζονται με το ελεγκτικό συνέδριο, την ανάγκη πιο λεπτομερών στοιχείων για τα οικονομικά μέσα. Θα ζητήσουμε ξανά από το ελεγκτικό συνέδριο να μας ε, δώσει στοιχεία για τη, και για τη διαχείριση ε, και βεβαίως για την επιστροφή χρημάτων όταν ολοκληρωθούν τα προγράμματα στον κοινωνικό προπολογισμό. Τέλος, υπάρχει ένα αίτημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, για χρηματοδότηση. Χρειάζονται περισσότερο προσωπικό. Εάν θεωρείτε ότι αυτή η συνεισφορά είναι χρήσιμη, εμείς συμφωνούμε να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια, 1,8 εκατομμύρια πιο συγκεκριμένα, ε, έτσι να προσθεθούν περίπου 15 θέσει εργασία, ε, να προσθεθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μια καλύτερη επιχειρησιακή ανάπτυξη της, του ελεγκτικού, του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, τον Νοέμβριο του 2020 θα αρχίσει να λειτουργεί και το σύστημα διαχείρισης των διαφορών υποθέσεων Αυτά ευχαριστώ. Να δώσω για το ΕΛΚΑ το λόγο στο σχέδιο συγητή, τον κύριο Νοβάκοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πράγματι μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά παίρνω το λόγο ως ε, φρέσκος εισηγητής, μόλις διορίστηκα. Δεύτερη θητεία μου στην Επιτροπή Έλεγχου του Περιπολισμού και χαίρομαι που επιστρέφω Ιδίω για μια πολύ σημαντική έκθεση που είναι τιμή να είμαι για αυτήν σκιώδη εισηγητής. Με εισηγήτρια την τέως ε, Επίτροπο για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Εμείς είμαστε εδώ οι καλύτεροι φίλοι των φορολογουμένων και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε. Δεν είναι βέβαια στι αρμοδιότητε τη επιτροπή, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να μα απασχολήσουν και πρέπει να τα αναφέρουμε σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Το πρώτο είναι οι επενδύσεις για την προστασία των συνόρων και την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος. Νομίζω ότι υπηρεσίε όπως η Ευρωπόλ θα πρέπει να στηριχθούν οικονομικά για να μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτά που τους ζητούμε. Επίσης έχουμε κάποιες καταστροφικές εξελίξεις σε κάποιους τομείς της οικονομίας. Έχουμε ε, το αυτό πυρετό ε, που οδηγεί σε απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων κεφαλών ε, το χείριο ζωικό κεφάλαιο σε πολλές χώρες και η Επιτροπή μας νομίζω μπορεί να στηρίξει. Βέβαια χαιρετίζω όλες τις προτάσεις της συναδελφού Κρέτσου και θα καταθέσω και εγώ τις δικές μου ιδέες Και φαντάζομαι και στις συνεδριάσεις ε, συνδελής θα καταφέρουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή. Ολυγέ Σαστέλ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κρέτσου μια πλήρη μεστή έκθεση με πολλές ενδιαφέρουσε προτάσεις όπως αναφέρθηκε η χρηματοοικονομική διαχείριση πώς θα βελτιώσουμε τις οικονομικές αυτές σχέσει και πώς θα βελτιώσουμε την, το προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και θα βελτιστοποιήσουμε τις επιδόσεις μεταξύ άλλων εξορθολογισμό των δικτών και των στόχων, αυτό που προτείνεται και το οποίο το έχουμε προτείνει βέβαια και κατά το παρελθόν. Και περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια. Φυσικά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει το παν για τη μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφηση. Παραδόξω, ε, εκτιμήσει πληρωμών και δυνατότητα απορρόφηση μπορούν να βελτιωθούν μόνο με αύξηση και με καλύτερη τεχνική υποστήριξη που η τάση είναι πτωτική, αλλά πρέπει να προσέξουμε το στοιχείο αυτό. Όπως αυτά που βλέπω στην τελευταία έκθεση σε σχέση με το ελεκτικό συνέδριο και τα χρηματοδοτικά μέσα. Συμφωνώ και σε αυτά που λέτε για τη μεταναστευτική κρίση και τη διαχείριση και θα πρέπει να γίνει διάκριση και να ξέρουμε τι χρειάζεται για την ανάπτυξη για εκρίζωση φτώχεια ε, και την ε, περάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οικονομικά να στηριχθούν αυτοί οι κλάδοι και για του στόχου και το συγκεκριμένο στόχο υποστήριξη του προγράμματο Δάφνη. Φυσικά και είμαστε υπέρ ε, γιατί θέλουμε να αντιμετωπιστεί η κακοποίηση των γυναικών, ιδίω στο σπίτι. Είναι κάτι που απαντά συχνότατα στην Ευρώπη, δυστυχώ. Επίσης, συμφωνώ να δοθούν ε, τα επαρκή μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από το τέλος του 2020. Ήδη λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε την προκοδότηση αυτής της υπηρεσίας. Ε, περιμένω βέβαια και τα νέα στοιχεία που θα συμπληρώσουν την έκθεση της ε, εισηγητρίας. Και διαρωτώ με μήπως η Επιτροπή μας, μπορούμε να δούμε και άλλες προτεραιότητες βέβαια, μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να συνοηθούμε ε, και να έχουμε μία παράγραφο στο κείμενο που ε, θα επιτρέψει να δώσουν και άλλες επιτροπές ε, προσοχή σε κάποια θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία τα συζητήσαμε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. για το οποίο είτε δεν υπάρχει πάντοτε σωστή χρηματοδότηση, είτε στο Συμβούλιο υπάρχουν περικοπές. Τα είπαμε αυτά. Και χθε τα λέγαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή μα, λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσε μέσα σε μια παράγραφα πέρα από τα τεχνικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, να προβάλλει εκ νέου τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης, ε, της κλιματικής πρόκλησης, καινοτομία, το πρόγραμμα Horizon 2020, απασχόληση των νέων και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το πώ μπορούμε να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για την ψηφιοποίηση της κοινωνίας και την τεχνολογική ανάπτυξη. Νομίζω ότι μπορούμε σε μια παράγραφο που θα ε, προσθεθεί στο ήδη υπάρχον κείμενο να αναφέρουμε όλους αυτούς τους στόχους. Και ιδίως έχοντας υπόψη ε, την αρνητική πινελιά που έκανε στον προπολογισμό το Συμβούλιο, που στερεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό κονδύλια, τα οποία θα χρειαζόντουσαν ε, γιατί μιλάμε για στόχους που έθεσε το ίδιο το Συμβούλιο. Τέλος πάντων τους ανήγγειλε τον τελευταίο καιρό και περικόπτει τα σχετικά κονδύλια. Τέλος πάντων θα ήθελα να μπει μια τέτοια παράγραφος ε, για να μιλήσουμε για τις θεματικές εγκάρσεις αυτές προτεραιότητες. Ευχαριστώ. <laughs> Νομίζω πως θα μας απασχολήσει και στο μέλλον ακόμα πιο έντονα το ζήτημα του, της ΕΠΟ. Υπάρχει προφανέστατα ένα θέμα υποχρηματοδότησης και το ξεκίνημά της δεν ήταν και το καλύτερο. Θα πρέπει να συζητήσουμε και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πάντα ε, υπεράσπιζε την ΕΠΟ, όμως ε, αρκετά κράτη-μέλη θέλουν να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που θεωρούμε εμείς αναγκαίο. Ας δούμε όμως ε, τι έχει κάνει ο Όλαφ, τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη και τότε θα καταλάβουμε ότι ο αριθμός είναι πραγματικά πολύ πολύ μικρός και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες είναι τρομακτικές. Δεν έχει γίνει εισαγγελική έρευνα, δεν έχει δοθεί συνέχεια στο ζήτημα τα... Ε, και όχι μόνο δεν προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα τα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε των κρατών μελών. Νομίζω πως σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και πραγματικά να πω ότι το, η διακίνηση ανθρώπων είναι από τα χειρότερα, πιο ε, απεχθή εγκλήματα. Και σίγουρα είναι επιζήμιο για τα οικονομικά συμφέροντα της ε, Ένωσης, ε, διότι τα αποτελέσματα της ε, παραοικονομίας επηρεάζουν αρνητικά τον προϋπολογισμό μας και την τσέπη του Ευρωπαίου φορολογούμενου μας περιορίζουν σημαντικά. Γι' αυτό λοιπόν ε, όντως θεωρώ πολύ σημαντικό το έργο. Ε, κύριε Κρούς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να προτείνω κάτι για το πρώτο σημείο της οικονομικής διαχείρισης. Βλέπω πως ε, γίνονται προσπάθειες για ε, περισσότερες δράσεις, όμως έχω δει από την εμπειρία μου μέχρι τώρα ότι τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στο μείον, είναι στο 0,4%. Ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώ αυτά τα συν και τα πλήν. Ε, Πολύ θέλει να αλλάξει να πάει στο, 0, στο μείον 0,6. Δεν το βλέπω καλό. Αυτά τα αρνητικά επιτόκια, τα οποία μετά ε, περνάνε στις τράπεζες, έχουν επιπτώσει στον προϋπολογισμό μας. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώ εμεί θα είμαστε σε θέση ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διαθέσουμε τα κονδύλια αυτά εφόσον πρέπει να περιμένουμε να κάνει τον κύκλο του ε, το χρήμα. Όταν ε, τα χρήματα βρίσκονται στην ε, τράπεζα και κάθονται, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα αρνητικά επιτόκια και δεν με το θεωρήσετε αμεληταίο το ποσό αυτό. διότι θα πρέπει να διαθέσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να καλύψουμε αυτά τα αρνητικά επιτόκια. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλύτερο να προσθεθεί και ένα άλλο σημείο το οποίο θα αναφέρει αυτά τα αρνητικά επιτόκια, ότι δηλαδή θα πρέπει να ασκείται κάποιος έλεγχος, να παρακολουθείτε η κατάσταση. Αυτό θα πρότεινα. Ευχαριστώ. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω σε αυτή την πρόταση. Ή θέλετε να κάνουμε άλλη συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Ωραία, ωραία, θα μεταφέρουμε το ερώτημά σας γραπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, γραπτή διαδικασία. Αλλά να ξέρετε πως δεν ε, παίρνουμε προκαταβολές ε, δισεκατομμυρίων, δεν είναι τόσο γενναιόρο δωρά τα κράτη-μέλη. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που κάνατε, η πρόταση, οπότε θα το μεταφέρουμε, διότι πρόκειται για μεγάλα ποσά. Και σίγουρα αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Λοιπόν, θα δούμε. Ναι, βλέπω το Συμβούλιο χαμογελά. Ωραία. Κύριε Πέξα, έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πραγματικά γιατί μας δίνει μια σωστή εικόνα για το πρόβλημα και έχει υποβάλει κάποιες πολύ καλές προτάσεις και ο άλλος ο το Renew επίσης ε, είπε σωστά πράγματα. Αυτό που θα πρέπει ίσως να υποθεί είναι πώς χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά χρειάζεται περισσότερο έλεγχο. και να μπορούμε να μετρήσουμε τελικά πώς δαπανούνται τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι έτσι τα αποτελέσματα θα είναι πιο ε, ενδιαφέροντα. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να προσθέσουμε και αυτήν την ε, παρατήρηση. Κύριε Χάουαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία που ήμουν πραγματικό μέλος στην Επιτροπή αυτή. Ήμουν και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση. Αυτή η γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τις πτυχές εκείνες που έχουν να κάνουν με την, τις εκθέσεις περί απόδοσης, ε, τους στόχους, τους δείκτες, ε, το νέο σετ δεκτών δικτών. Ε, πρέπει να αναπτύξουμε, να, τα αναπτύξουμε περαιτέρω αυτά, ε, διότι έτσι γίνεται σωστός δημοσιονομικός προγραμματισμός. Συμφωνώ με την κυρία Κρέτου ε, η οποία με την εμπειρία της σίγουρα θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Τώρα για τα trust funds. Ακούστε, στην Επιτροπή αυτή υπάρχει ένα ζήτημα διαφάνειας του προπολογισμού της Ένωσης σε όλες τις πτυχές του. Τα trust fund παίζουν ένα ρόλο, βεβαίως έχουν ένα σκοπό, ένα λόγο ύπαρξης, αλλά πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη διαφάνεια και υπάρχουν και άλλες πτυχές της, της διαφάνειας του προπολογισμού που θα είναι ε, θα αποτελούν όλο, όλο και μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Εγώ όταν ξεκίνησα ε, δεν ήθελα καθόλου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που αρχίζει από B, ε, μάλλον το Brexit εννοεί ο μιλητής. Πάντως η συνεισφορά στα έστωτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το εξωτερικό θα πρέπει να είναι σίγουρα πιο διαφανής. Και αυτό θα αποτελεί πρόκληση καθώς θα περνάει ο καιρός. Και ένα τελευταίο σημείο στα πλαίσια της υπηρεσίας δεν είναι μόνο το θέμα του, του, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και καιρό στη Μοσυνομική Επιτροπή και νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας και αυτή την Επιτροπή. Ε, μια υπηρεσία, η Frontex, ε, οδηγείται σε πολύ σημαντική αύξηση του προπολογισμού της τα επόμενα χρόνια. Πέρα από το 2020. Εάν δούμε πώς αυξάνονται οι δαπάνες, ε, ακόμα και το 2019, η επέκταση διεύρυνση Frontex που έχει κατά νου η Κομισιόν θα, θα, θα αποτελέσει μια τεράστια πρόκληση ε, για την υπηρεσία αυτή, για τις διαχειριστικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν. Ε, θα πρότεινα λοιπόν η Επιτροπή αυτή να δώσει μεγάλη προσοχή στην επέκταση αυτής ε, της υπηρεσίας, στην διεύρυνσή της, στην πρώτη φάση διεύρυνσης για να μπορέσει αυτό το εγχείρημα να στεφθεί από επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ καλή παρέμβαση. Το είδαμε, τα είδαμε στην ΕΑΣΟ σήμερα. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε ικανοποιημένοι. φυσικά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι μαζί σας, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας την έκθεσή σας. Θα ήθελα μόνο να κάνω δύο-τρία σχόλια για την έκθεση. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε δώσει το Κοινοβούλιο μία έκθεση ε, για τις μακροπρόθεσμες ε, εισρωές και εκροές. Ε, αρχές Ιουνίου εγκρίθηκε αυτή η έκθεση και είμαστε διατεθειμένοι να σας το στείλουμε εκ νέου εφόσον χάθηκε. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις αναφορές μας ε, για την απόδοση. Δεν, είναι μόνο, δεν έχουμε μόνο τις δηλώσεις προγραμματικές, ε, έχουμε και μικρές περιλήψεις του προγραμμάτων που περιγράφουν τι κάνει το πρόγραμμα και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Σε ό,τι αφορά τώρα την βελτίωση, σε ό,τι αφορά τις αναφορές και τις εκθέσεις, και, και για τα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή ενώση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, αυτό αφορά και τους τον αριθμό των δικτών, συνδέεται ε, με τη ε, διαδικασία που ακολουθείται στα πλαίσια του νέου MFF, του νέου πολιτικού Θα δούμε λοιπόν πώς θα εκδηθούν τα νέα προγράμματα για το επόμενο πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό θα θα κρίνει πολλά. Υπάρχει έκθεση για τη μετανάστευση που είναι όσο γίνεται πιο πλήρης. Ε, βεβαίως δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε τις δαπάνες του μεταναστευτικού τομέα. Θα σας στείλουμε σε αυτή την έκθεση εφόσον δεν είναι διαθέσιμη ε, στα μέλη ε, της, του Κοινοβουλίου για τον Ντάφνε, πολύ σημαντικό πρόγραμμα. του δίνουμε πολύ, πολύ μεγάλη σημασία Νομίζω το έχουμε πει και στα τα προηγούμενα χρόνια. Εμεί δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική δημοσιονομική γραμμή γι' αυτό. Το πρόγραμμα αυτό τη χάνει καλή προώθηση. Υπάρχουν σημαντικά ποσά στα ετήσια προγράμματα εργασιών. Σε ό,τι αφορά την, ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Κομισιόν δεσμεύεται για τη δημιουργία αυτή τη υπηρεσία και να αρχίσει να λειτουργεί όπω προβλέπεται στα τέλη του 2020. Έχουμε αξιολογήσει τι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το 2020 και στην πρόταση προϋπολογισμού για το επόμενο έτος οι δεσμεύσεις είναι υψηλότερες ε, από ό,τι είχαν προβλεφθεί αρχικά ε, στο ε, στις νομοθετικές δηλώσεις. Θα τα ξαναδούμε βεβαίως όλα αυτά και θα προβούμε σε τροποποιήσεις εφόσον χρειαστεί. Θέλουμε οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε πιο διαφανείς και όλο και καλύτεροι στο μέτρο του δυνατού. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now I pass the floor to our rapporteur, Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγητρία μας, την κυρία Κρέτσου. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω, εσάς ε, κυρία Πρόεδρε και τη Γραμματεία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Νοβάκοφ με μεγάλη χαρά ε, συνεργάστηκα μαζί του για την έκθεση αυτή και όπως είπα και στην αρχή λίγα στοιχεία μόλις ε, σας παρουσίασα ε, τα οποία σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις που νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα προσαρμοστήκαμε σε δύσκολους καιρούς, χρειάστηκε να δαπανίσουμε χρήματα για τη Frontex και άλλα σχετικά. Είναι η πρώτη φορά που ζητήθηκε από την Ένωση να χρηματοδοτήσει τη διαχείριση συνόρων. Επίσης, είχαμε έρευνα και καινοτομία σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, πράγματα που θέλουμε να προωθήσουμε. Είμαι πράγματι τέος επιτροπός, άρα γνωρίζω πολύ καλά από τότε που ήμουν στη Ρέτζη τι θα πει έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Έτσι θα διευκολύνουμε τη ζωή των δικαιούχων των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται με το δέοντα τρόπο. και προς όφελος των πολιτών πάνω απ' όλα. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ήρθα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της κακής διαχείρισης των χρημάτων των φορολογουμένων. Πολύπλοκη έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι κατέθεσαν τις συστάσεις και προτάσεις τους και μαζί με τη γραμματεία της Επιτροπής θα συνεχίσω να μελετώ όλα αυτά τα σημεία. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο εφόσον ε, είναι πολλές οι γενικές διευθύνσεις ε, μονάδες ε, που επιλαμβάνονται και επειδή διατέλεσα επίτροπος γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα αλλά για ζητήματα όπως είναι το Ντάφνη και άλλα προγράμματα, νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο για να συνεργαστούμε μαζί με την Κομισιόν και να καταλήξουμε σε ένα ξεχωριστό κονδύλι για το Ντάφνη. Σίγουρα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη του πληθυσμού από τη βία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Πρόεδρο. Ευχαριστώ όλους θα ήταν εδώ σήμερα και ελπίζω συντονισμένα να μπορέσουμε να εργαστούμε. Γιατί είναι πλοκό το σχέδιο της έκθεσης αυτής. Είναι και πολλές άλλες επιτροπές που συμμετέχουν και το γεγονός ότι Πρέπει να λάβουν υπόψη και τις δικές τους τοποθετήσεις. Προκλήσεις υπάρχουν και είναι πολλές. Το 2020 πρέπει πλέον να έχουμε αναπτύξει τη ταχύτητα. Έχουμε την πρόκληση της μετανάστευσης αλλά και άλλα θέματα όπως για παράδειγμα πώς θα προετοιμαστούμε για το 2020, για να προχωρήσουμε περαιτέρω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αν δεν εκριθεί και το προσεχές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027 θα έχουμε Πολλού κινδύνου να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Επίσης πρέπει να ξαναρχίσουν ε, οι τριμερεί διάλογοι, οι οργανικές διαπραγματεύσει για αυτό το πιδελταπή. Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη αυτή έκθεση. Περιμένουμε ανυπομονησία τι τροπολογίε. Έχω όμως και ένα δυσάρεστο καθήκον να πρέπει να διορθώσω την ημερομηνία για την προθεσία, προθεσμία καταστροπολογιών. Δεν είναι η δεκάτη, αλλά η ενάτη η Σεπτεμβρίου. Είχα πει δύο, θα πω τέσσερις το μεσημέρι, για να έχετε λίγο παραπάνω ώρα. Βέβαια, το κοινοβούλ... Ε, η γραμματεία μας θα είναι πολύ χαρούμενη ε, να πάρει έως το νωρίτερα τις τροπολογίες. Ε, θέλω να την κυρία Κρέτσου. Και λέω ότι 9 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία που ισχύει και στις προηγούμενες τρεις εκθέσεις που συζητήσαμε. Να καλωσορίσω την ομάδα του Όλαφ Χαιρόμαστε που μας επισκέπτεστε. Να καλωσορίσω όλους ιδιαίτερα στο Γενικό Διευθυντή. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Ήδη μας απασχόλει υπόθεση Άσο. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί στην Επιτροπή Ελεκτού Προϋπολογισμού και ε, με βάση μάλιστα τα πορίσματα μιας έκθεσης δικής σας σχετικά. Να δώσω το λόγο μας στον πρόεδρο για να κάνει την ομιλία του, να μας κάνει την παρουσίαση και έπειτα... Α, μπορούμε να δούμε, βλέπω και στην οθόνη της διαφάνειές σας. Λοιπόν, κύριε Ήταλα, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. And Ευχαριστώ, κυρία, κυρία Πρόεδρε, Εξότιμα μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και σας συναντώ και σας παρουσιάζω βεβαίως την ε, εκδοχή του 2018 της έκθεσης της Όλαφ. Το 2018 ο Όλαφ ε, συνέχισε την ε, έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο ελέγχου με δύσκολες, περίπλοκες, ευρεία κλίμακας έρευνες ανά την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Μέσω των συστάσεων της, ο Όλαφ, του, Όλαφ εξασφαλίζει ότι τα χρήματα τα ευρωπαϊκά τα οποία δεν τα πανήθηκαν με τον σωστό τρόπο θα ανακτηθούν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το 2018 ο Όλαφ ε, εξέδωσε 256 συστάσεις στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και ανέκτησε, μάλλον σύστησε την ανάκτηση 371 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω αυτής της δουλειάς έρευνας ο Όλαφ αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και προστατεύει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από την απάτη. Είναι μια κρίσιμη υπηρεσία που προσφέρει όλα στους Ευρωπαίους πολίτες. Για μας είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως εσείς, αλλά και οι πολίτες, να αντιληφθούν την ουσία του ερευνητικού έργου του Όλαφ και τις πρόσφατες τάσεις που έχουν φέρει στο φως οι έρευνές μας. Βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι ένας πλήρης κατάλογος ολοκληρωμένων ερευνών, όμως ε, ο υπερεθνικός χαρακτήρας των εργασιών του όλα του δίνει την ευκαιρία να έχει μια πιο πλήρη εικόνα των αλλαγών, των εναλλασσόμενων τάσεων της απάτης ανά την Ευρώπη. Το 2018 είχαμε μεταξύ άλλων σε επίπεδο ελέγχου διασνοριακά ε, συστήματα απάτης όπου εικονικές εταιρείες χρησιμοποιούνται για να κρύβουν ε, ψεύτικες εμπορικές συναλλαγές. Αποφυγή τελωνιακών δασμών από οργανωμένο έγκλημα. Απάτη κατά την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωρικών προϊόντων. Οργανωμένο έγκλημα και, και ε, συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος σε ό,τι αφορά κονδύλια που χρηματοδοτούν κανονικά κέντρα προσφύγων. Θα δώσω κάποια πρακτικά παραδείγματα σήμερα για να σας δείξω πώς ο Όλαφ προστατεύει την ασφάλεια και την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών, πώς η αναλυτική δυνατότητα του Όλαφ στον τομέα των τελωνίων είναι μοναδική και πρέπει να ενισχυθεί, πώς η πραγματογνωμοσύνη του Όλαφ που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία 20 χρόνια είναι κρίσιμη για να επιληθούν περίπλοκες δυσμιουργικές υποθέσεις και πως ο Όλαφ έχει αναπτύξει μια μοναδική δυνατότητα έρευνας σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Για το πρώτο σημείο πρώτα, ο Όλαφ παίζει έναν ρόλο κλειδί ως ένας κόμβος γνώσεων και συντονισμού συνδέοντας τις εθνικές τελωνιακές αρχές ανά τον κόσμο. Ήμασταν εξαιρετικά ενεργοί το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια καταπολεμώντας ε, τα, το εμπόριο, το παραεμπόριο μάλλον παραπημένων προϊόντων. Αυτή, αυτό το λαθρεμπόριο ε, προκαλεί ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία και βεβαίως υπονομεύει τις ε, νόμιμες επιχειρήσεις και διακυβεύει την απασχόληση. Τα παραπημένα προϊόντα είναι μια τεράστια, έχει ένα τεράστιο τζίρο και έχουμε επικεντρωθεί έχουμε κεντρώσει τι προσπάθειές μας σε προϊόντα που εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία μας, το περιβάλλον όπως ε, το ε, παραπημένο σαμπουάν, ε, τα εξατήματα αυτοκινήτων ή ακόμα και τρόφιμα τα οποία έχουν παραπηθεί. Να δώσω πρώτα ένα παράδειγμα. Το πρώτο παράδειγμα είναι το, το σαμπουάν. Είναι πολύ αγαπημένο προϊόν για τους απαταιώνες, διότι μπορεί να πουλήσει κανείς εκατομμύρια μικρά μπουκαλάκια σε χαμηλές τιμές ανά τον κόσμο. Το 2018 λάβαμε πληροφορίες ε, για την εξάρθρωση μιας παράνομης, ενός παράνομου εργοστασίου στην Κίνα που παρήγαγε παραποιημένο σαμπουάν. Το τελευταίο, η τελευταία αποστολή είχε ήδη φύγει από το εργοστάσιο και επειδή η Ευρώπη ήταν πιθανό να είναι ο προορισμός, αρχίσαμε να παρακολουθούμε τη διαδρομή αυτού ε, του φορτίου. Ήταν περίπλοκη η διαδρομή του, πέρασε από διάφορα λιμάνια στην Κίνα, στην Κορέα, στο Μεξικό, στην Κολομβία. Όταν οι ερευνητές του Όλαφ εκτίμησαν ότι αυτό το παραπημένο σαμπουάν μπορεί ε, και κινδύνευε μάλλον να εξαφανιστεί πριν φτάσει στον προορισμό του, ο Όλαφ ειδοποίησε τις αρχές της Κολομβίας και του Μεξικού και 400 τόνοι παραποιημένου σαμπουάν με μια αξία λιανικής πώλησης 5 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν σε συνεργασία με τις Ισπανικές και Αμερικανικές αρχές. Τα τελευταία χρόνια ο Όλαφ καταπολεμεί επίσης μια άλλη μορφή απάτης εξαιρετικά επικερδή που είναι η υποεκτίμηση των κλωστεφατοργικών ε, και προϊόντων και των υποδημάτων που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τελωνίων ε, σε πολλά κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σλοβακία, στην Τσεχία αλλά και στην Ελλάδα. Τα αγαθά από την Κίνα φτάνουν σε κοντέινερ πάνω σε πλοία που συνήθως μπαίνουν στην Ευρώπη από το λιμάνι του Αμβούργου. Τα κοντέινερ τα οποία θεωρητικά είναι σε τράνζιτ, στη συνέχεια φορτώνονται σε φορτηγά και μεταφέρονται για, τελωνια... για εκτελονισμό κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί οι εγκληματίες θεωρούσαν ότι μπορούσαν να δηλώσουν πολύ χαμηλές ε, πλαστές, πλαστές χαμηλές αξίες. Η τελευταία περίπτωση αφορά ε, εισαγωγέ κλωστοφοντουργικών και υποδημάτων στην Ελλάδα από το 2015 στο 2018. Με βάση τα ευρήματα, το Όλαφ έκανε μια σύσταση οικονομική προς τα ελληνικά τελωνία για να ανακτήσουν 202 εκατομμύρια ευρώ τελωνιακών δασμών που είχαν χαθεί. Ο Όλαφ έστειλε επίσης μια δικαστική σύσταση ε, στην, ε, στην εισαγγελία καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η έκτη τέτοια υπόθεση του Όλαφ που ολοκληρώθηκε από το 2016. Σε αυτές τις έξι υποθέσεις συνολικά ο Όλαφ έχει κάνει οικονομικές συστάσεις για πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό των ε, τελωνιακών δασμών που δεν πληρώθηκαν και διέφυγαν του ευρωπαϊκού, του Βεβαίω, οι εκτιμόμενε απώλειες σε επίπεδο ΦΠΑ είναι ακόμα μεγαλύτερε. Εδώ, σε αυτέ τι περιπτώσεις, όλα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να ε, προλάβει αυτή την απάτη και την απώλεια εισοδημάτων. Και βεβαίω να και βοηθάει ταυτόχρονα τι εθνικέ τελωνιακέ αρχέ στο έργο του. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να διευρύνουμε τι δυνατότητέ μα να εργαστούμε ε, ω ένα κέντρο ανάλυση στοιχείων τελωνιακών για να ενισχύσουμε έτσι και την Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση με βάση και τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Βόντερ Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές του Όλαφ έχουν επίσης αντιμετωπίσει ε, αύξηση ενός συγκεκριμένου τύπου ε, ε, απάτης. Απάτη κατά την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Παραδείγματο χάρη ο Όλαφ ολοκλήρωσε μια σειρά από έρευνε όπου οι ίδιοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια σε μια σειρά από project που αφορούν την προώθηση των ευρωπαϊκών κρατικομικών προϊόντων. Οι δράστες προσέγγιζαν εμπορικά επιμελητήρια στα κράτη-μέλη και πρόσφεραν βοήθεια ε, λέγοντας ότι θα, θα μπορέσουν να βρουν ασφαλή ευρωπαϊκά κονδύλια και θα δώσουν πρακτική υποστήριξη για την εφαρμογή των project. Όταν εγκρινόταν τα project, ήταν η στιγμή ε, οι απαταιώνες να πάρουν τα χρήματα. Για να το κάνουν αυτό, δημιουργούσαν μια σειρά από εικονικές επιχειρήσεις που έπαιζαν το ρόλο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαχωνισμό, των προμηθευτών και των αρχών ε, ε, εφαρμογής αυτές οι υπηρεσίες δεν είχαν πουθενά ούτε έδρα, ούτε εργαζόμενους, απλά ανέβασαν, φούσκωναν τις τιμές για τις υπηρεσίες που ορισμένε φορές ούτε καν υπήρχε παροχή υπηρεσιών αυτών. Στη συνέχεια υπήρχε ξέφλημα χρήματο μέσω τραπεζικών λογαριασμών στην Ευρώπη αλλά και τρίτες χώρες όπως η Ουκρανία και οι παρθένες νήσοι τη Βρετανία. Ο Όλαφ έκανε πάνω από 30 επιτόπιους ελέγχους σε διάφορα κράτη-μέλη. Μίλησε με μάρτυρες και ανέλησε ε, στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα και οδηγήθηκε σε μια οικονομική σύσταση προς την Τζιάγκρη για την ανάκτηση 7,7 εκατομμυρίων ευρώ και να προλάβει την δαπάνη άλλων 7,3 εκατομμυρίων ευρώ με δικαστικές συστάσεις προς ε, την εισαγγελία των Βρυξελών αλλά και της Σόφιας. Να μια περίπτωση που πραγματικά χρειάζεται 20 χρόνια εμπειρία ε, κατά πολέμηση της απάτης για να μπορέσει να διδουκανθεί. Το 2018 ο Όλαφ ολοκλήρωσε μια σειρά από υποθέσεις που είχαν να κάνουν την εξωτερική βοήθεια όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για έρευνα εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία από τις υποθέσεις αυτές. Στην υπόθεση αυτή, ο Όλαφ ανακάλυψε ότι μια Ιταλική εταιρεία είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών που τη βοηθούσαν να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν σχέση με διαδικασίες προμηθειών αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία. Η Ιταλική αυτή εταιρεία δωροδόκησε επίσης υψηλόβαθμους αξιωματούχους έτσι ώστε να επηρεάσει την, αξιολόγηση, την Επιτροπή Αξιολόγησης που τελικά έδινε ε, την σύμβαση στην Ιταλική εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Όλαφ συνεργάστηκε στενά με την εισαγγελία της Βορείας της Μακεδονίας, την εισαγγελία του Μιλάνο καθώς και την Guardia di Finanza, την Ιταλική ε, Οικονομική Αστυνομία, η Όλαφ. Ε, ο Όλαφ ε, έκανε μια σειρά από συνεντεύξεις μαρτύρων και επιτόπιους ελέγχους, καθώς ε, και επιχειρήσεις για την εξέβρεση υλικού δαχτυλικών αποτυπωμάτων στην έδρα της εταιρείας. Ο Όλαφ αυτό το συμπέρασμα και στην σύσταση στην οικονομική προς την Engineer για την ανάκτηση του συνόλου του ποσού που είχε διατεθεί. Επίσης υπάρχει δικαστική ε, σύσταση προς τις ταλικές αρχές για να προβούν σε δίωξη των εν λόγω ατόμων. Επίσης, Όλα βεβαίως ζήτησε αυτή η Ιταλική εταιρεία να μπει σε μια μαύρη λίστα για να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας επίσης ξεκίνησαν από την πλευρά του μία ε, έρευνα ποινικού περιεχομένου. Όπως γνωρίζετε, όλα φέχει και εντολή να ερευνά ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Προσωπικού υπάλληλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει την φήμη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Όπω και άλλοι εργοδότε, έτσι και τα ευρωπαϊκά όργανα κινδυνεύουν από την απάτη που να προέρχεται από το δικό του προσωπικό σε σχέση με την αμοιβή του, σε σχέση με τι δαπάνε του, Κινδυνεύουν επίσης από τη διαφθορά. Το 2018 ο Όλαφ ολοκλήρωσε 27 έρευνε για σοβαρέ παρατυπίες ε, και λανθασμένες συμπεριφορέ ε, ε, υπαλλήλων της Ένωσης, 17 των οποίων οδήγησαν σε συστάσεις. Στον τομέα των ιστορικών αυτών ερευνών το 2018 ο Όλαφ ασχολήθηκε με έναν σημαντικό αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με ευρωπαϊκές υπηρεσίες καθώς και με αντιπροσωπείες σε τρίτες χώρες. Όπως άλλωστε συζητήθηκε νωρίτερα. Και τώρα θα εξετάσουμε τη συνεργασία του, του Όλαφ με τους εταίρους του και τη σημαντική συμμετοχή του στην ανάπτυξη των πολιτικών καταπολέμησης της διαφθοράς. Η απόφαση δημιουργίας της ΕΠΟ αποτέλεσε ορόσημο στην ε, προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Όλα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την ΕΠΟ έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων προστατεύονται από την απάτη και τη διαφθορά και, στην, ε, και στα συμμετέχοντα και στα μη συμμετέχοντα κρατημέλη. σε όλο το 2018 ο ΛΑΦ συνεργάστηκε ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εκτελεστική της υπηρεσία για την αναθεώρηση της ε, στρατηγικής της ε, Κομισιόν κατά της απάτης και συντόνισε την εφαρμογή της. Η λοιπόν στρατηγική υιοθετήθηκε το 2019, η οποία προτείνει μεταξύ άλλων ε, ανάλυση δεδομένων για την ε, καταπολέμηση της απάτης. Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, βλέπετε οι υποθέσεις μας δεν είναι καθόλου εύκολες. Πολύ συχνά είναι αρκετά περίπλοκες και για να μπούμε στην ουσία του προβλήματος χρειαζόμαστε συνεργασία με τους εταίρους μας. Τώρα, ως ε, νέος Γενικός Διευθυντής ε, του Όλαφ έχω τρεις ε, βασικές αρχές οι οποίες διέπουν η... πρώτα απ' όλα η διαφάνεια, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη. Για την εμπιστοσύνη όμως προϋπόθεση είναι οι άλλες δύο. Μέχρι, από το διορισμό μου μέχρι τώρα έχω συναντηθεί με διάφορους φορείς, με την Ευρωπόλ, τη Euro, το Συμβούλιο, το Ελεκτικό Συνέδριο και άλλους φορείς και φυσικά τις αρχές των κρατών μελών. Την ίδια προσέγγιση θέλω να χρησιμοποιήσω για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλω η ΕΠΟ, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να είναι ένα εγχείρημα που θα στεφτεί με επιτυχία. Και την πρώτη ε, στιγμή που θα έχω τη δυνατότητα θα ασχοληθώ με προσοχή με την ΕΠΟ. Όμως, ε, ας δούμε λίγο τις ε, τάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι σαν τη γάτα με το ποντίκι. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ το συντονισμό ε, των εθνικών αρχών και των ε, τελωνιακών αρχών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με καλύτερο τρόπο. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει κάποιος που θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες, όλη τη γνώση για να μπορούν να χρησιμοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι όλα ε, διαθέτει τόσο το προσωπικό όσο και την εμπειρογνωμοσύνη για κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη. Αν η εμπιστοσύνη υπάρχει, τότε μπορούμε να λάβουμε τη γνώση από τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και να τη χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν υπάρχει η γνώση, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και στη συνέχεια να επιστρέψουμε ε, το, την ε, γνώση αυτή στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις τις οποίες αν αναλύσουμε με προσοχή και αξιολογήσουμε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δύο κυρίαρχες τάσεις είναι απάτη τροφίμων και περιβαλλοντική. Ο οργανισμός μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ε, καταπολέμηση της απάτης, ιδιαίτερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πιστεύω πως ε, ειδικά αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους πολίτες και όλα είναι εδώ για τα συμφέροντα των ε, πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γενική Διευθυντή για την εξαιρετική παρουσίαση η οποία μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή εικόνα ε, του τι κάνει όλα και το επιτελείο σας και να ξέρετε πως εκτιμούμε πάρα πολύ το έργο σας. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια ή η Βιόλα έχει ζητήσει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Διευθυντή, για την παρουσίαση της έκθεσης και για τις ε, λεπτομέρειες που μας παρουσιάσατε. Είμαι καινούργια Ευρωβουλευτής και καινούργιο μέλος της Επιτροπής. Γι' αυτό εξεπλάγει όταν έλαβα την έκθεσή σας ε, λιγότερο από μία ημέρα πριν την ε, συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συνήθεια εδώ, αλλά αν θέλετε να γίνει ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτά που κάνετε, νομίζω πως θα ήταν καλό να μας δίνατε την ε, έκθεση νωρίτερα. Είχατε αρκετό χρόνο για να βρείτε έναν τρόπο, νομίζω, να μεταδώσετε την πληροφορία. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας συστήσω, τουλάχιστον για το επόμενο έτος, να βρείτε κάποιον τρόπο για να μας ε, διαβάσετε τις πληροφορίες αυτές νωρίτερα, εγκαίρως. Έπειτα, αναφερθήκατε σε ορισμένες ε, περιπτώσεις που εξετάσατε σε ορισμένε υποθέσεις που εντυπωσιάζουν μεν στο χαρτί, αλλά όπως έχει ήδη γίνει συζήτηση και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αγγελία, όταν η υπόθεση αυτή περνάει από εσά στα χέρια των εθνικών αρχών, δηλαδή στο, στα κράτη-μέλη, αλλάζει τελείω η αντιμετώπιση. Το κάθε κράτο μέλο την χειρίζεται διαφορετικά. Έχετε λοιπόν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για το πώ τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν και χειρίζονται τις υποθέσεις που τους περνάτε. Έχετε δηλαδή στοιχεία για το αν συνεχίζουν οι έρευνες μετά, σε τι ποσοστό, αν ε, υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν ποιο κρατός μέλος συνέχισε τις έρευνες και ποιο όχι και για ποιους λόγους. Ασκείτε εσείς ε, κάποια πίεση στα κρατημέλη. Από αυτά που διάβασα, είναι κάπως λυπηρό ότι ο εισαγγελέα ε, πάγωσε την υπόθεση Μπάμπης δεν ξέρω λοιπόν αν εμεί σε αυτή την Επιτροπή θα μπορούσαμε να στηρίξουμε το έργο σας ε, κάπως περισσότερο και να ασκήσουμε πίεση στον ε, εισαγγελέα. Ο κύριος Μπάμπης ε, δεν είναι... είναι και πρωθυπουργό, ξέρετε. Δεν είναι ένα απλό πολιτή. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε αν υπάρχει κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε, να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο έτσι ώστε να βοηθήσουμε. Θεωρείτε πως όταν κατονομάζουμε κάποιον έχει ουσιαστικό όφελος, πως ασκείται, θα ασκηθεί, ας πούμε, στην περίπτωση του κύριου Μπάμπης, πολιτική πίεση. Υπάρχει κάποιος τρόπος να σας βοηθήσουμε. Κυρία Μπένκοβα. Έχετε το λόγο, κυρία Μπένκοβα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ιταλά. Δύο σύντομες ερωτήσεις στα βουλγαρικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση και τις πολύ αναλυτικές πληροφορίες που μας δώσατε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου πριν, στην έκθεση αυτή μας αναφέρετε πολλές υποθέσεις ε, απάτης που ερευνήσατε στα κράτη-μέλη και αναφέρατε και μία υπόθεση που αφορά δική μου χώρα, τη δική μου χώρα ε, και απάτη με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες όμως για τις εταιρείε και για τη δράση που αναλαμβάνεται σε βάρος ε, των απαταιώνων. Τι μέτρα έχετε λάβει ποιες είναι οι συνέπειες για τους απατεώνες αυτούς. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι που αναφέρατε στη δική σας την παρουσίαση. Πριν από κανένα χρόνο περίπου είπε όλα αυτά ότι θα υπάρξει ένα σύστημα πληροφοριών για την αποτροπή απάτης με τα κοινοτικά κονδύλια. Πώς προχωρά αυτό το σύστημα πληροφοριών. Υπάρχει κάποια δημόσια πληροφόρηση επ' αυτού. ευχαριστώ. κύριε Κατερίνα Κινίτσι τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστώ την Ριοϊτάλα για την πολύ χρήσιμη παρουσίαση αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις που μας δίνουν και μια ιδέα νομίζω για το πόσο πολύπλοκο είναι το έργο του Όλαφ. Εξίσου δύσκολο είναι να διωχθούν οι δράστες ε, των ε, οικονομικών αυτών εγκλημάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή, να ευχαριστήσω και το προσωπικό σας. Ένα σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω από την έκθεση που κάνατε και το οποίο αφορά το οργανωμένο έγκλημα. και συγκεκριμένα για τα εγκλήματα σε βάρος των οικονομικών σφαιρών της Ένωσης. Είπατε ότι εστιάζει εκεί όλα μεταξύ άλλων. Σίγουρα πρέπει να το προσέξουμε και μιλήσατε για τη συνεργασία του Όλαφ με τη Eurojust αλλά και το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι αυτό κομβικό ε, στο πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας με τα διάφορα θεσμικά όργανα. Και σε σχέση με ένα προηγούμενο ερώτημα να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, συζητούμε την ε, αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού. Και θα έχουμε και το θέμα του κανόνα παραδεκτού. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι ανοιχτό ακόμη. Και όλα αυτά πάντα υπό το πρίσμα του έργου σας για την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας. Η κυρία Κάταλιν Τσέχ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ταλά, η τέτοια έκθεση για το 2018 είναι, δίνει μια πολύ γλαφυρή εικόνα, θετική για τις έρευνες, για τις επιτυχίες σας και όλα αυτά είναι ευχάριστα και σας συγχαίρω. Από την άλλη πλευρά όμως, Υπάρχει ακόμη πολλά, υπάρχουν ερωτηματικά ε, για τη διαφθορά και τις σχετικές μελέτες που δείχνουν ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Θα μπορούσατε να έχετε κάνει περισσότερη προσπάθεια για να εντοπίσετε τέτοιες περιπτώσεις και να δείτε αν υπάρχει συστημικός χαρακτήρας, π.χ. στα καταπιστευματικά ταμεία ή αλλού. Ούτε στην πράξη, ούτε στη θεωρία βλέπουμε και πολλά να κάνει όλα αυτά, αλλά ούτε και κομισιόν για την αντιμετώπιση αυτών των συστημικών προβλημάτων. Για την προστασία των χρηματοπιστωτικών συμφερόντων. Καλό θα ήταν η συμμετοχή στην εισαγγελία να είναι προϋπόθεση για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτά για την Κομισιόν και προς τον κύριο Ήταλα. Συμφωνείτε πως ε, όλα αυτά πρέπει να κάνει ενδελεχή ανάλυση για να δει κατά πόσο υπάρχουν απειλές συστημικού χαρακτήρα για τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Ένωσης και αν υπάρχει τέτοιο συστημικό κίνδυνο, είστε υπέρ του να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα θέματα στην ετήσια έκθεση του όλα. Δεύτερον, δυστυχώ, πολύ λίγη πληροφόρηση υπάρχει ε, για το τι γίνεται μετά από τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Τι κάνετε πέραν της αναφοράς, ε, πέραν της υποβολής εκθέσεων, ε, για να υπάρχει μια συνέχεια, μια διαδικασία που θα παρακολουθεί και θα βλέπει κατά πόσο μετά τις ε, συστάσεις υπήρξαν και κάποιες καταδίκες ή καταγγελίες. Και τι γίνεται όταν ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες είτε ε, επαγγελθούν κατηγορίες ή όχι, σίγουρα υπάρχουν και κανόνες προστασία δεδομένων, αλλά υπάρχει κάποια δημοσιοποίηση των υποθέσεων και τι κάνει η Κομισιόν ή η Όλαφ οι εκθέσεις τη Όλαφ να θεωρούνται ε, τεκμήρια από τις ε, ποινικέ αρχές τη Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουαρτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Γενικό Διευθυντή για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και εξαιρετικά διαφωτιστική. Είναι πιο εύκολο να κάποιος ε, ε έχει απέναντί του τον ε, συνομιλητή του. Έχω κάτι, κάποια απλά και απευθείας ερωτήματα να στείλω, ευθεία ερωτήματα να σας ε, κάνω. Πρώτα απ' όλα, ο όγκος ε, για την ανάκτηση που συστήνεται. Είναι μια οργάνωση 60 εκατομμυρίων. Εσείς συστήνετε 371 εκατομμύρια ευρώ προς ανάκτηση. Το 2017 ήταν 3,9 δις. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διακυμάνσεις. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι πόσα από αυτά τα χρήματα τελικά ανακτώνται. Καλό είναι, καλή είναι η σύσταση, αλλά τα χρήματα αυτά τελικά όντως επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με την οργάνωσή σας. Ποιες είναι οι, οι πιο σημαντικές δημοσιονομικές ε, πιέσεις που νιώθετε στη δουλειά σας. Και τρίτον, και είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα, Ποια είναι η άποψή σας για το συνολικό επίπεδο της απάτης στην Ευρώπη. Αυξάνεται ή μειώνεται. Ο κύριος Μικούλας Πέ, Πέτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω τσεχικά. Δύο ερωτήματα έχω να θέσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξέρω εάν αληθεύει ότι ότι υπάρχει μια υποστήριξη από το 2018 για μια υπόθεση για την οποία, την οποία σταματήσατε να την, μελετείτε, να την, να την διερευνείτε. Είναι ένα σκάνδαλο που σταματήσατε να εξετάζετε αυτή την υπόθεση και να κρατήσουμε να να χρησιμοποιήσει τελικά τα κονδύλια αυτά. Πρέπει να προλέπτουν κυρώσεις. Δεν μπορούμε να γνωρούμε τέτοιες υποθέσεις. Η κυρία Αγγέλικα Βίντσιχ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. κατά τη διάρκεια του προεκλογικού μα της προεκλογικής μας εκστρατείας ε, είχαμε πολλές ερωτήσεις από πολίτες ακριβώς για αυτά τα θέματα, για θέματα απάτης και μάλιστα κάποιος ε, με ρώτησε για μία περίπτωση ενός ε, φοροτεχνικού που κάλυψε διάφορες απάτες, γεωργικές απάτες που είχαν να κάνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια. δεν, ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Ναι. Νομίζω πως είναι δική μας ευθύνη και καθήκον ως ευρωβουλευτές να ενημερώνουμε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Σαντο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γενικό Διευθυντή για αυτή την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Όλαφ. Όπως είπατε και εσείς, είναι προς το συμφέρον όλων μας να χρησιμοποιούμε ε, με τρόπο χρηστό τα χρήματα των φορολογούμενων προς όφελός τους. Η διαφθορά γιγαντώθηκε στην Ουγγαρία, έγινε κομμάτι της καθημερινότητας στη χώρα ε, κυρίως λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση. Και νομίζω πως αυτά που άκουσα επιβεβαιώνουν αυτές τις απόψεις. Και εγώ πραγματικά ντρέπομαι που ακούω τέτοιες περιπτώσεις. Η καταχρήση στην Ουγγαρία μεταξύ του 2014 και 2018 είχαν οδηγήσει στον Όλαφ να αποκαλύψει περιπτώσεις όπου τεράστια ποσά υπεξαιρέθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω αν μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα παραπάνω για αυτά τα νούμερα που βλέπω εδώ και τι γίνεται, πώς ε, αντιμετωπίζετε αυτές τις περιπτώσεις. Τι βήματα μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να αντιστραφεί αυτή η τάση στο μέλλον. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις μήπως για εμάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νοβάκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Ιτάλα για τις προσπάθειες του και για τη δουλειά του. Θυμάμαι την ακρόαση του πέρυσι όταν ήταν υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Νομίζω πως αρκετοί συνάδελφοι και εγώ ανάμεσά τους είχαμε αναποθέσει αποθέσει τις ελπίδες μας στην ετοιμότητά του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Νομίζω πως έχει κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Αλλά να δούμε λίγο, λίγο πιο προσεκτικά τα νούμερα. Πριν από τρία χρόνια περίπου Είχε γίνει μια συζήτηση για το γεγονός ότι όλα αφανίγει πολλές έρευνες, αλλά τις κλείνει χωρίς σύσταση. Και θυμάμαι μάλιστα μια περίπτωση όπου ήταν 70-80 υποθέσεις ανοιχτές για ένα πρωί μόνο. Επίσης, έχετε εκδώσει 256 συστάσεις. Πόσες από αυτές ε, έχουν ακολουθήσει τα κρατημέλη. Και οι υποθέσεις απάτης που ξεσκεπάσατε, κατά πόσο επανορθώνεται η ζημιά, κατά πόσο επιστρέφουν τα χρήματα αυτά που υπεξαιρέθηκαν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. μπορούμε να συζητάμε ώρες, μέρες για αυτά τα θέματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τις εθνικές, τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να διεξάγονται έρευνες. Για να αποδοθούν και ευθύνε. Όταν κάποιος κάνει κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν νομίζετε πως έχει έρθει ο καιρός ε, για να ασκεί αυτόνομα όλα αυτά τις δικές του έρευνες έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει ε, περισσότερες ε, υποθέσεις, να συνεργάζεται για παράδειγμα με τις εισαγγελίες, με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας ε, συγχαρώ. Είμαστε και συνάδελφοι άλλωστε από παλιά. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Την πρώτη ήδη έγινε θα ήθελα να την επαναλάβω. Όλα συντάσσει αιτήσιες εκθέσεις και σε αυτές τις αιτήσιες εκθέσεις ε, δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ε, συστάσεις. Κάνει, κάνει μάλλον συστάσεις. και για κυρώσεις σε ορισμένες ε, προβληματικές, ιδιαίτερα προβληματικές περιπτώσεις. Επίσης υπάρχουν κονδύλια που έχουν ε, υπεξαιρεθεί και πρέπει να επιστραφούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις ε, για να λύσει το πρόβλημα αυτό, για να βελτιωθεί η κατάσταση, επηρεάζονται τα κονδύλια για τη συνοχή, για παράδειγμα, για τις ε, περιφέρειες. Από την άλλη, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις, τι αποφάσεις είναι αυτές και τι αφορούν. αν για παράδειγμα Όλαφ κάνει μια σύσταση που αφορά μεγάλα ποσά, 370 εκατομμύρια ευρώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς αντιδρά. Δεύτερη ερώτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείται η αντιπολίτευση της Ουγγαρίας, βέβαια, αλλά θεωρώ ότι προσπαθούν έτσι με την ανοιχτή κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας ε, να μπαλώσουν λίγο τα πράγματα για το, για το άσχημο εκλογικό αποτέλεσμα. Προσπαθούν δηλαδή λίγο να ρίξουν στάχτη στα μάτια για να ανέβουν εκείνοι. Μας είπατε ότι διεξάγονται 18 νέες έρευνες για υποθέσεις ε, που σε, στο σύνολό τους είναι λιγότερες από ότι το, την τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, έχουν ακουστεί αρκετά για συστάσεις και τις συστάσεις που κάνει ο Όλαφ συστάσεις που αφορούν τα κονδύλια που, δι, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουγγαρία. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες συστάσεις για μείωση του ποσού από 3,5 έως ε, και πάνω από 5%. Εγώ όμω θέλω να ρωτήσω κάτι που ίσως δεν τολμούν να ρωτήσουν άλλοι. Κύριε Γενική Διευθυντή, υπάρχει μήπως κάποιο συστημικό πρόβλημα στην χρήση, στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ουγγαρία ή όχι, διότι η αντιπολίτευση της Ουγγαρίας λέει ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Έτσι όμως όπως το βλέπω εγώ, ο Λαφ δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο σημασία το αν το πρόβλημα είναι συστημικό ή όχι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Όμως θα ήθελα να μου απαντήσετε για το αν θεωρείτε εσείς πως το πρόβλημα είναι συστημικό ή όχι. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Κύριε Ήταλα, παρακαλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα τα οποία ήταν πολλά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω και για όλες τις ερωτήσεις. Όπως είπατε είναι τόσο πολλές ερωτήσεις ε, που ενδεχομένως να ξεχάσω κάποια. Θα κάνω ό,τι μπορώ και μπορούμε να επανέλθουμε ενδεχομένως αργότερα. Ξεκινώντας από την έκθεση του Όλαφ που τη λάβατε χθες. Τη λάβατε χθες γιατί δημοσίευθηκε χθες. Ίσως του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα Ήταν λίγο περίεργο το χρονοδιάγραμμα αυτή τη φορά. συνήθω τον Ιούλιο δημοσιεύουμε την έκθεση, αλλά λόγω των εκλογών πήγαμε πιο πίσω. Πάντω το σημειώσαμε. Θα το συζητήσουμε και με την γραμματεία σα για το πώ μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Ρωτήσατε ε, πώ μπορούμε εμεί να πιέσουμε πολιτικά ε, κάποιον ο οποίος ε, διώκεται. Δεν είναι δική μας δουλειά κάνουμε να ισχύσουν πολιτική πίεση. Εμεί κάνουμε την έρευνα. Συντάσσουμε την έκθεση, την στέλνουμε στις αρχές και οι αρχές αποφασίζουν τι θα κάνουν. Αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει πολλές φορές. Ότι πρέπει να πάμε λέει παραπέρα. Αλλά εμεί έχουμε ένα κανονισμό πολύ συγκεκριμένο. Ε, και έχουμε καθήκοντα πολύ συγκεκριμένα. Και αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, ε, Ερωτήσεις για το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν κάποιες τάσεις που δείχνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι όλο και πιο δημιουργικό, όλο και πιο περίπλοκο και πρέπει πάντα εμείς να τρέχουμε από πίσω. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ε, πόσα προσόντα έχουν οι, οι ερευνητές μας εδώ μιλάμε για τον κανονισμό, για αυτό, ενώ δεν έχουμε καν πρόσβαση ε, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η εταιρεία, το οργανωμένο έλλειμμα οργανώνει με οργανώνεται με εικονικέ εταιρείε ε, σε διάφορε χώρε όχι μόνο τη Ένωση, αλλά και εκτό Ένωση. Ε, αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί, είναι και στα χέρια σα να μα δώσετε τα εργαλεία για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί διότι η εγκληματίας ε, είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από μας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πως είναι κοινός στόχος όλων να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Τώρα, ε, για τον κανονισμό. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι έχουμε συζητήσει και το Κοινοβούλιο έχει πάρει θέση, το προηγούμενο τουλάχιστον Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τους επιτόπιους ελέγχους και βεβαίως το ΦΠΑ. Και εκεί το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε τις θέσεις της Όλαφ και ελπίζω να βρεθεί μια λύση και στο Συμβούλιο για να φτάσουμε σε έναν καλό κανονισμό γρήγορα. Πάντως είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για μας, για τη δουλειά μας. Τώρα, τι συμβαίνει μετά τις έρευνές μας και τι γίνεται με τις συστάσεις μας. Αυτό το ρώτησαν πολλοί. Να προσπαθήσω να το διευκρινίσω. Όταν διεξάγουμε την έρευνά μας, αυτή η έρευνα είναι διοικητικού τύπου. Στη συνέχεια βεβαίως παραδίδουμε την έκθεση στις εθνικές αρχές ή στην εισαγγελία μιας χώρας παραδείγματος χάρη. Αλλά η στην εισαγγελια μια χωρας παραδειγματο χαρη αλλα η δικη μας δουλειά τελειώνει με την έκθεση. Δεν είμαστε εμείς το όργανο που θα ανακτήσει τα χρήματα. Είχαμε μια συζήτηση και το χειμώνα με την έκθεση ΕΓΚΑΦ, τελικά πόσα ανακτάτε. Δεν είναι δική μα δουλειά. Δεν κάνουμε εμεί την ανάκτηση των χρημάτων. Βεβαίω θέλουμε να βοηθήσουμε για την ανάκτηση. Από εκεί πέρα όμω, ε, άλλε υπηρεσίε τη Επιτροπή είναι υπεύθυνε γι' αυτό. Και εφόσον γίνει κατανοητό αυτό, σίγουρα υπάρχει υπερθωριό βελτίωση τη ανάκτηση. Ε, η Κομισιόν έχει αρχίσει να το εξετάζει πιο προσεκτικά το θέμα αυτό και έχει δημιουργηθεί ένα Corporate Management Board ε, στην ε, ε, Κομισιόν, υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Budget, υπάρχει η Όλαφ, ο Γενικός Διευθυντής και κάθε φορά που κάνουμε μία σύσταση οι άλλες Γενικές Διευθυντήσεις πρέπει να απαντήσουν για το τι έκαναν με την ανάκτηση αυτή. Και τότε αυτό το όργανο, το Corporate, Corporate Management Board, τα ελέγχει όλα αυτά. Βεβαίω είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με να πούμε ότι η τάδε σύσταση οδήγησε σε τόσα, τόση ανάκτηση φέτος. Διότι η ανάκτηση μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια, σε δέκα χρόνια. Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε δηλαδή το τι προτείνουμε εμεί με την πραγματική ανάκτηση, διότι η ανάκτηση λαμβάνει χώρα αργότερα. Πάντως ε, υπάρχει συνεργασία με τις άλλε γενικέ διευθύνσει και ψάχνουμε το σωστό τρόπο. Τώρα, οι δικαστικές συστάσεις τέθηκε το ερώτημα του ε, προς ποιε χώρες έχουμε συστάσεις ε, και τι έγινε μετά. Είναι 41 υποθέσεις, μπορείτε να τι δείτε μία προ μία. Έγινε και ένα ερώτημα για την Ουγγαρία. γενικότερα να πω ότι βεβαίως όταν βλέπουμε τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και συζητούμε με τις αρχές των κρατών Όμως τα στοιχεία δεν είναι πάντα σωστά. Πρέπει κανείς να κοιτάξει πίσω από τα στοιχεία για να δει την πραγματική κατάσταση στην κάθε χώρα όπως και να έχουν τα πράγματα, εγώ έχω αποφασίσει να εξετάσω όλα τα κράτη-μέλη, να συναντήσω τις αρχές τους και αν χρειαστεί και αν το θελήσουν και τα κρατη ε, να συναντήσω και τους πολιτικούς θύνοντες ε, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γιατί είναι τόσο χαμηλό, λέμε, το ποσοστό καταδίκης. Ε, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία. Πριν από μερικούς μήνες ε, ήμουν στην Βουλγαρία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση εκεί με την εισαγγελία και μας εξήγησαν διότι ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό ε, καταδίκης και μας είπαν είναι τόσο δύσκολο με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τις παρατυπίες εκεί ε, σε σχέση με το δικό μας ποινικό κώδικα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις αριστοιχίες. και αποφασίσαμε, διότι του στείλαμε μια υπόθεση ε, και μια έκθεση, αποφασίσαμε να έχουμε ένα σημείο επαφής. Όταν υπάρχει μια υπόθεση που αφορά τη χώρα αυτή, πάμε στην εισαγγελία και προσπαθούμε να εξηγήσουμε από κοντά για το τι πρέπει να γίνει. Αυτοί βέβαια γνωρίζουν καλύτερα το εθνικό τους ποινικό δίκαιο και ξέρουν από εκεί πέρα τι να κάνουν. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και με τις προσωπικές επαφές, αν θέλετε. Έγινε ένα σεμινάριο, ένα κογκρέσο με τους εθνικούς εισαγγελείς τον Ιούλιο και έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Εξετάσαμε τις διάφορες, διάφορες πραγματικές υποθέσεις και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. και πήγε πολύ καλά αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικαστικές ε, ε, συστάσεις, βεβαίως εδώ θα βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σαν τους λόγους ε, ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όποιος και αν είναι ο κανονισμός, και βεβαίως είναι πολλά τα εκκρεμή ζητήματα για το ποια μορφή θα πάρει ο κανονισμός, Όταν θα έχουμε τον νέο κανονισμό, ελπίζω να είναι όσο γίνεται καλύτερο. Αλλά η άλλη μια φορά είναι θέμα συνεργασίας. Θέλω να μπορώ να πάω στο Λουξεμβούργο να συναντήσω τον εισαγγελέα και να δούμε υπόθεση πώς ξεκινάει η συνεργασία. Να μπορούμε να έρθουμε εδώ και να πούμε ξέρετε συνεργαστήκαμε για το θέμα, για το τάδε θέμα και είχαμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι σημαντικό για τον Όλαφ, να δείξουμε ότι έχουμε διάθεση συνεργασίας. Τώρα είναι πολλά τα εκκρεμή ζητήματα. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε όταν θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τέθηκε και ένα ερώτημα για το stock farming, για την ε, κτηνοτροφία. Νομίζω ότι εδώ υπήρξε μια παρανόηση σε φορά κάποια νέα που κυκλοφόρησαν σήμερα για μια υπόθεση. Όταν ερευνούμε, διερευνούμε μια υπόθεση, πάντα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση με κοινοτικά χρήματα. Εάν ικανό, όμως το κράτος μέλος έχει μεταφέρει τα χρήματα αυτά σε άλλο project, τότε το συγκεκριμένο project πλέον είναι, αφορά μόνο εθνικά χρήματα. Οπότε δεν είναι δική μα αρμοδιότητα πια το θέμα. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε αν δεν αφορά κοινοτικά χρήματα. Αυτό προβλέπει ο κανονισμό για την ώρα. Τώρα τέθηκε και ένα ερώτημα για την ενημέρωση των πολιτών για αυτά που κάνει ο Όλαφ. Είναι σημαντικό αυτό. Σας είπα ότι μια από τις βασικές αρχές για μένα είναι διαφάνεια. Πρέπει να είμαστε διαφανείς και προσπαθούμε να πούμε περισσότερα για αυτά που κάνουμε. Όμω ε, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία. Ακόμα και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ε, υποθέσεις εν εξελίξη. Είναι εμπιστευτικέ. Η διαφάνεια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για εκκρεμεί υποθέσεις. Όταν ολοκληρωθεί βεβαίως η υπόθεση, κάποια στιγμή ακόμα και ο εισαγγελέα έρχεται και εξηγεί την υπόθεση στο κοινό. Μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Και διαφάνεια σημαίνει ότι ξέρετε τι κάνει ο Όλαφ, γνωρίζετε αυτές τις τάσεις και μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαντήσουμε. Και έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εμπιστοσύνη, να, ξέρουν, να ξέρει και ο κόσμος τι κάνει ο Όλαφ. Διότι πολλά χρόνια τώρα ακούω από το Κοινοβούλιο ότι δεν ξέρουμε τι κάνει ο Όλαφ. Εμεί προσπαθούμε να ερχόμαστε εδώ όσο γίνεται πιο συχνά. Για να σα εξηγήσουμε τι κάνουμε. Πάντω σίγουρα θέλουμε να βελτιώσουμε το θέμα της επικοινωνίας, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι πολίτες, πώς να έρθουν σε επαφή με τον Όλαφ. Το ίδιο ισχύει και με του εμπλεκόμενους φορεί Ε, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν μα βοηθούν στι υποθέσει. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μας, ε, μας ε, έρχονται σε εμά με υποθέσεις. Μας τις αναθέτουν. Ναι, τώρα τα αποδεικτικά στοιχεία και το κατά πόσο είναι παραδεκτά. Είναι εξαιρετικά προβληματικό αυτό. Και για τα αριθμητικά στοιχεία, διότι όταν υποβάλλουμε μια έκθεση και ε, τα στοιχεία αυτά δεν είναι παραδεκτά στο δικαστήριο είναι πρόβλημα. Η Κομισιόν στο νέο κανονισμό προτείνει να είναι παραδεκτά σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές υποθέσεις. Αυτό ήδη βοηθάει κάπως. Ήταν δύσκολο βέβαια, διότι πολλές φορές εμείς δίνουμε τα στοιχεία, η Εθνική Εισαγγελία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ξεκινάει από την αρχή και έτσι χάνεται χρόνος. Τώρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα να βληθούν κάπως. Ήταν πολλές ερωτήσεις. Τα πρακτικά προβλήματα σε πλευρά εσόδων ε, και το θέμα αυτό της, της ε, Το είχαμε πει ήδη στην προηγούμενη έκθεση, πέρυσι, στη μεγάλη εκείνη υπόθεση. Τώρα συνεχίζεται. Είναι μια τάση, είναι συστηματικό πλέον. Πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό με τα εθνικά τελωνία. Και Χρειαζόμαστε και καλύτερα εργαλεία ε, για την ανάλυση δεδομένων και τη χρήση των πληροφοριών. Έτσι είναι αυτά. Μετά είχαμε το ερώτημα των φετινών στοιχείων και των περσινών. Αυτό σχετίζεται άμεσα με αυτή την υπόθεση της υποεκτίμησης, διότι αυτή η υπόθεση του Μένου Βασιλείου ήταν τεράστια. Μιλάμε για δύο δισεκατομμύρια τώρα δεν είχαμε τέτοια υπόθεση φέτος. Αυτό από μόνο του εξηγεί την απόκληση. Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ωραία. Προσπάθησα να απαντήσω σε όσο γίνεται προς ερωτήματα. Σίγουρα θα ξέχασα κάτι. Μπορώ να επανέλθω πάντως και διμερός. Θέλω να σας συναντήσω όλους και προσωπικά. Έτσι δεν να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε τα ζητήματα, διότι σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος. Και θέλω να καλέσω την Επιτροπή σας στα... στις εγκαταστάσεις του Όλαφ, στα γραφεία μας και μπορούν να σας εξηγήσουν εδώ οι διευθυντές μας το τι κάνουμε. Είστε καλοδεχούμενοι που σου βρείτε χρόνο να έρθετε στα γραφεία μας. Να βρούμε μια μέρα που να σας βολεύει και εσάς για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Και βεβαίως ε, και για το μέλλον του Όλαφ να συζητήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιταλά. Σας ευχαριστούμε και για την προθυμία σας και για την πρόσκληση που μας απευθύνετε να επισκεφθούμε τα γραφεία σας. Θα διαβιβάσω την πρόσκληση στην Πρόεδρο για να τη συζητήσουμε. Και προχωρούμε με το τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης, ε, ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων ε, του Επιτροπής εποπτείας ε, του ΟΛΑΦ για το 2018, πρόεδρος ο κύριος Γιάν Μούλντερ. Έχετε το λόγο κύριε Μούλτερ και αν κάποιος από τους ε, συναδέλφους σας θέλει το λόγο, ευχαρίστω στη συνέχεια. Εσείς παρακαλώ κύριε Μούλτερ. Thank ε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι καταρχάς θα σας εξηγήσω τη γενική τάση, τις γενικές τάσεις και Ραφαέλα, ο συνάδελφος, θα σας, ε, ο Ραφαέλ Μουνιός θα σας πει κάποια πιο συγκεκριμένα ε, στοιχεία για το 2018. Η Επιτροπή Εποπτείας σημειώνει ότι το 2018 ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών. Νέος Γενικός Διευθυντής, που με τον ορισμό του είχαμε κι εμείς ε, συμμετάσχει στην όλη διαδικασία από πριν. Εκδώσαμε μια γνωμοδότηση για να δούμε κατά πόσον ικανοποιητικά ολοκληρώθηκε η δικασία πρόσληψης και πράγματι αυτό συνέβη και κάναμε και μια θετική σύσταση. Έχουμε με την άφηξη του νέου Γενικού Διευθυντού μια νέα εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Μπορεί κάποιοι να γνωρίζετε τις προηγούμενες εκθέσεις της Επιτροπής Εποπτείας. Σε αυτές τις προηγούμενες εκθέσεις πάντα υπήρχε ε, μία ε, ένταση ε, μεταξύ των δύο, δηλαδή Γενικού Διευθυντού και Επιτροπής Εποπτείας. Αυτό δεν θα το βρείτε αυτή τη φορά. Σίγουρα μπορεί να έχουμε διαφωνίες κάποιες φορές, αλλά η σχέση μας είναι πολύ καλή. Και το εργασιακό περιβάλλον αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Το δεύτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή Εποπτείας ήταν ότι το 2018 είχαμε πολλές απουσίες στη γραμματεία. Ήταν πολύ αναρωτικοί, άλλοι μεταφέρθηκαν, ε, μετατέθηκαν σε άλλη υπηρεσία κτλ. Άρα κάναμε λιγότερα από αυτά που είχαμε προβλέψει στην αρχή του έτους. Χρειάστηκε να περιοριστούμε μόνο σε όσα υπαγορεύει ο κανονισμός. Να δώσουμε δηλαδή όπως πάντοτε βέβαια ειδική και ιδιαίτερη προσοχή σε διαδικασίες, τη διάρκεια των ερευνών, και να συμφωνήσουμε με το σύστημα αναφοράς. Θέλει βελτιώσεις ακόμα, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από ό,τι πριν. Επίσης, ένα θέμα ήταν η βελτίωση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τακτικά επισκεπτόμεθα το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προσπαθούμε να έχουμε στο ένα καλύτερο συντονισμό. Και αν γίνει και η ανταλλαγή αυτή προσωπικού θα έχουμε ένα μέλος από το ελεγκτικό συνέδριο στην Επιτροπή Υποπτείας του Όλου. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς θα γίνει, αλλά έχουμε μεγάλες προσδοκίες και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Η Κομισιόν επίσης προτείνει ένα νέο κανονισμό να αναθεωρηθεί ο κανονισμός δηλαδή 883 και η Επιτροπή Υποπτείας παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις. και θα σας διαβιβάσουμε και σε σας και στο Συμβούλιο συστάσεις. Ήδη περιλαμβάνει πρόταση κάποια πράγματα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα λοιπά. Άλλα πράγματα τα οποία επισημαίνουμε είναι αυτές οι εκθέσεις 12 μηνών και τι θέλουμε να ισχύει και δικαίωμα πρόσβαση στι πληροφορίε είναι ένα ειδικό όρο, μια προπόθεση. Κατά το παρελθόν, ζητούσαμε πληροφορίε από του προηγούμενου γενικού διευθυντέ. Και μα λέγανε, ναι, ναι, ωραίο το ερώτημα, αλλά δεν σα αφορά το θέμα. Αυτό το θεωρούμε παράδειγμα σε Επιτροπή Εποπτεία. Αν λοιπόν θέλουμε εμεί να λάβουμε κάποια πληροφορία που θεωρούμε απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας, θα πρέπει να μπορούμε να την έχουμε. Θα κάνουμε τη σχετική σύσταση. Επίσης, η θέση της γραμματείας είναι ένα άλλο θέμα. Ανήκε στην Όλαφ μέχρι πριν τρία χρόνια. Όπως είπα όμως, οι σχέσεις μεταξύ γραμματείας και διευθυντού της Όλαφ δεν ήταν οι βέλτιστες δυνατές. Γι' αυτό αποφασίστηκε η γραμματεία να είναι εκτός Όλαφ. στο τμήμα προσωπικού της Κομισιόν μεταφέρθηκε. Περίπου τρία χρόνια είναι που έχει γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας που να είναι ικανοποιημένο με αυτή την εξέλιξη. Άρα μια άλλη σύστασή μας είναι να το ξαναδούμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Να βγουν τρεις λέξεις δηλαδή από τον κανονισμό. Εκτός του Όλαφ όπου θέλει στην Κομισιόν, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Επιτροπή Εποπτείας χαίρεται ιδιαίτερα από σχεδόν όλες οι συστάσεις που κάναμε στην προηγούμενη Επιτροπή, γιατί τώρα στην διαφορετική έγιναν αποδεκτές. Και εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν στην τελική συνεδρίαση στην Επιτροπή με μεγάλη πλειοψηφία. Ελπίζω και στον επερχόμενο τρομερή διάλογο οι απόψει και οι γνωμοδοτήσει αυτές της επιτροπή εποπιά θα επιβιώσουν και θα περιληφθούν στον νέο κανονισμό. Αυτή τη στιγμή εξεργαζόμαστε εκθέσεις για την κατάσταση προσωπικού στην Επιτροπή Εποπτείας που βελτιώνεται με ταχύ ρυθμού. και ελπίζουμε στα τέλη του έτου, να είμαστε πλήρω τελεχωμένοι οπότε να προχωρήσουμε με άλλες εκθέσεις για τις dismissed cases όπως τις λέμε και άλλες υποθέσεις που θα μας απασχολήσουν. Και σε σχέση με τη συζήτηση που προηγήθηκε. Να πω ότι και εμείς ως Επιτροπή ανησυχούμε ιδιαίτερα με το τι γίνεται, με το ποια συνέχεια έχουν οι συστάσεις του όλα ότι δεν είναι ικανοποιητικό να εργάζεται πάνω σε μια υπόθεση όλα, να υποβάλει συστάσεις στο κράτος μέλος και να λέει ευχαριστούμε αλλά δεν θα πάρουμε. Να μην κάνει τίποτα. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Θα, θα σας υποβάλουμε σχετική αναφορά επ' αυτού. κάτι το παρελθόν. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας ιδίω με την πρόεδρο, την Ίνκεμπορ Γκρέσλε, την πρώτη τη προηγούμενη θητεία. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί με την επιτροπή αυτή, υπό την τη σύνθεση η καλή αυτή συνεργασία. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Ραφαέλ Μουνιώθ, ο οποίο θα σα αναφέρει κάποιε άλλε πτυχέ τη έκθεση. Καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι για πρώτη φορά στην Επιτροπή σα για την ανταλλαγή αυτή απόψεων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΟΛΑΦ. Όπω γνωρίζετε, ο λόγο ύπαρξή τη Επιτροπή Εποπτεία ε, είναι ακριβώ ε, η παγρύπνηση της, για την ανεξαρτησία του Όλαφ. Γι' αυτό και θέλουμε να, είναι, να ρυθμίσουμε ακριβώ τον τρόπο με τον οποίο προχωρά στις έρευνε τη. Θέλουμε να υπάρχει όμω και διοικητική και δημοσιονομική αυτονομία του Όλαφ, γιατί αυτή η ανεξαρτησία έχει άμεση επίπτωση και στο πώς ολοκληρώνονται οι έρευνες. Λαμβάνοντας υπόψη σήμερα τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα ήθελα να εστιάσω στην δημοσιονομική αυτή πτυχή που εμείς ως Επιτροπή Εποπτείας αναφέρουμε στην πεπραγμένων μας με τον τίτλο «Έλεγχος των πόρων που έχει του Όλαφ» και συγκεκριμένα μιλάω για τις παραγραφους παραγράφους από 9-33. Η Επιτροπή Εποπτείας θεωρεί πως η ανεξαρτησία ιδιοσιονομική του ΟΛΑΦ έχει άμεση επίπτωση στην αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων και ερευνών της. Θεωρούμε σημαντικό λοιπόν ο προπολογισμό αυτός να είναι επαρκής, να είναι δεδειγμένος, αλλά και η στρατηγική των ανθρωπίνων πόρων να είναι ολοκληρωμένη. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρούμε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να πρέπει να εφαρμόσει όλα τα αυστηρά μέτρα εξοικονόμηση σπόρων που εφαρμόζονται από τις άλλες γενικές διευθύνσεις κομισιών. Ίσα ίσα που θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα που θα ευνοούν την πρόσληψη άκρως εξειδικευμένου και ικανότατου προσωπικού για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη τις μελλοντικές σχέσεις εργασίας Όλαφ και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Επιτροπή Εποπτείας στηρίζει την ειδική μεταχείριση της Όλαφ και αυτό σημαίνει, από οικονομικής πλευράς πάντα, σημαίνει ότι θα απαιτείται και η μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση των κονδυλίων από τον Όλαφ. Και τώρα θέλω να σας αναφέρω μέσα από τις ανησυχίες μας στην Επιτροπή Εποπτείας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το κομμάτι του προπολογισμού που αφορά τη θρομολόγηση του... της βάσης δεδομένων για τη διαχείριση περιεχομένου, OCM. για τα εργαλεία και την ε, και τις ευθύνε και τις ε, αρμοδιότητες παρακολούθησης και ελέγχου που θα έχει όλο. Αυτό λοιπόν το σύστημα πληροφορικής για τη διαχείριση των ε, του περιεχομένου είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Γιατί αν δεν λειτουργήσει σωστά θα επηρέασει αρνητικά την καθημερινή εργασία των ερευνητών, της ε, υπηρεσία. Όπως ήδη έγινε σε μια περίπτωση και έχει περάσει και τη δική μα δουλειά. Αν δούμε τις, τα ερωτηματολόγια για την ικανοποίηση του προσωπικού, βλέπουμε να μειώνονται τα ποσοστά με τη δρομολόγηση και εφαρμογή του συστήματος αυτού διαχείρισης περιεχομένου το SM στα αγγλικά. Αν και το 2018 κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση. Γιατί είναι η ερώτηση. Γιατί μας ανησυχεί η διαχείριση αυτού του συστήματος, του περιεχομένου. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι επηρεάζει τη λειτουργία, το λειτουργήμα, αν θέλετε, ε, του ερευνητή, που είναι ίσως το σημαντικότερο στο πλαίσιο του ΟΛΕΦ. Επίσης, μας απασχολεί γιατί η ευρή ανταλλαγή πληροφοριών και σε σχέση και με το τι προβλέπεται στο μέλλον με τη συνεργασία της ΟΛΑΦ και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ε, που θα αυξήσει την επιχειρησιακή δυνατότητα του ε, συστήματος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος OSM και μας απασχολεί και το κόστος αυτού του project. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λάβει διαφορετικές εκτιμήσεις κόστους, όλο και προς τα πάνω. Τελικά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το οριστικό κόστος αυτού του έργου, άπαξ και όλα πληρωθεί. Στην γνωμοδότηση παριθμών 1 2018, η Επιτροπή Εποπτείας συνέστησε σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου τη διενέργεια ελέγχου για τα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει στο ΕΣΥΕΜ από το 2012. Οπότε και αποφασίστηκε να αναπτυχθεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή, να περιληφθεί εκεί το αίτησιο κόστος, στην παράγραφο 26 δε της γνωμοδότησης για το προπολογισμό στην γνωμοδότηση 1 του 2019, η Επιτροπή Εποπτείας ε, συστήνει εκ νέου. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του OCM να γίνει μια πλήρης ε, επισκόπηση της διαδικασίας για να οριστούν ε, οι διάφορες ευθύνες των διαφόρων που συμμετείχαν. Το Δεκέμβριο του 2018 το σύστημα διαχείρισης περιεχομένων που πολλές φορές έχω πει, το SEM τέλο πάντων στα αγγλικά, έχει μια νέα δομή διακυβέρνησης. Έχουμε την διευθύνουσα επιτροπή, έχουμε τον πρώτο, τον νέο γενικό διευθυντή, που καθορίζει τις απαιτήσεις του νέου συστήματος σε ό,τι τη ροή εργασία. Έχει οριστεί ξεκάθαρα πλέον. Και από ό,τι φαίνεται στην πράξη λειτουργεί καλά. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, γιατί δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, είναι ότι μία από τις ε, αρμοδιότητές μας είναι η έρευνα σε σχέση με τη διάρκεια των ερευνών της Όλαφ. Λέμε στην έκθεσή μας ότι σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την ποιότητα των εκθέσεων που βάλει όλα αυτά στην Επιτροπή Αποπτίας για τις υποθέσεις με πάνω από 12 μήνες διάρκεια, οι περισσότερες εκθέσεις δεν περιλάμβαναν ουσιαστικές πληροφορίες ό,τι αφορά την περιγραφή της υπόθεσης, ώστε η Επιτροπή Αποπτίας να μπορέσει να αξιολογήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα όλα και αν είναι κατάλληλα αυτά τα μέτρα. Τέλο, καταλήγουμε στην έκθεσή μα ότι η ποιότητα των πληροφοριών δεν έχει βελτιωθεί σε ό,τι το συγκεκριμένο ε, πάντοτε θέμα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Επίσης, στην παράγραφο 49 της ε, έκθεσή μα αναφέρουμε πώς θα πρέπει να λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας έχοντας υπόψη ότι το καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε τα τρία θεσμικά όργανα για το έργο της όλα, Συμβούλιο, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, που άλλωστε μας έχουν εκλέξει και έχουν ορίσει και τα μέλη μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος Επιτροπής, φαίνεται να βελτιώνονται οι σχέσεις με την ε, εκλογή του νέου Γενικού Διευθυντή του Όλαφ, δεν έχουν αυτούς τους μήνες που έχουν παρέλθει, επιληφθεί το αντίθετο μάλλον τα προβλήματα που είχαμε διαπιστώσει κατά το παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελε κάποιος ευρωβουλευτής να πάρει το λόγο για αυτά που μόλις ακούσαμε. Νομίζω πως σιγά σιγά φαίνεται η κούραση σε όλους μας. Όποιος όμως έχει ακόμα κουράγιο μπορεί να λάβει το λόγο, μπορεί να μείνει εδώ και να σχολιάσει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από τον Όλαφ. Αγαπητέ Πέτρη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι, στη μετάφραση άκουσα κούραση. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει κούραση. Με συγχωρείτε που άρχισα να γυρίσω ή έπρεπε να πάω σε μια άλλη επιτροπή ταυτόχρονα ε, όπου πάλι είχε γίνει παρουσίαση της ε, Προεδρίας. Θα κάνω λοιπόν μερικά σχόλια ή ερωτήσεις που θα παρουσιάσω τώρα. Γνωρίζω τις ε, περιστάσεις που αναφέρθηκαν και κάποιες από αυτές μου κάναν ιδιαίτερη εντύπωση. Στην έκθεση δραστηριοτήτων, στην ε, παράγραφο 68, αναφέρεται ότι η Επιτροπή τονίζει τη σημασία που έχει ο Όλαφ να αναλάβει πρωτοβουλίε στον εντοπισμό και ανάλυση κινδύνων απάτη ε, που θα βασίζεται στην τακτική ανταλλαγή πληροφοριών με τι άλλε γενικέ διευθύνσει. Για κάποιον που δεν ξέρει την κατάσταση, αυτό θα τον θα εκπλήξει. Ε, γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κανονικά θα έπρεπε. Αυτό φυσικά το λέω σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει από, τον, ε, από τις έρευνες, το τι δηλαδή ερευνάτε και τι όχι. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Μάλντερ να μου πει λίγα λόγια παραπάνω για αυτά τα ευρήματα και για τις συστάσεις τις οποίες δεν θεωρώ πολύ λογικές. Κατά τα άλλα βλέπω μια αρκετά έντονη γλώσσα. Να σας πω και ακριβώς πού. Στην απάντηση του νέου Γενικού Διευθυντή στις συστάσεις που διατυπώσατε ε, θεωρείτε ότι δεν τις έλαβε καθόλου υπόψη σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στην έκθεση δραστηριοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι αν θα μπορούσατε να επεκταθείτε και να μας πείτε τι εννοείται. Ωραία, θεωρώ λοιπόν πως ε, ο κύριος Σαβαρμα ήταν ο τελευταίος που τοποθετήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα, τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Μάλντερ να απαντήσει και να κάνει τα καταληκτικά του σχόλια. Κύριος Μόλτερ, Γιάν. Ωραία λοιπόν, θα λάβω πρώτος το λόγο σε ό,τι αφορά την παράγραφο 69. Ναι, νομίζω πως δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Τα λόγια τα εξηγούν όλα από μόνα τους. Δεν καταλαβαίνω εσείς τι πρόβλημα έχετε, διότι τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στις δραστηριότητες του Όλαφ. Είναι μια κάπως γενική δήλωση και δεν νομίζω ότι υπονοεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συστάσεις του Γενικού Διευθυντή, εγώ δεν αναφέρθηκα σε συστάσεις της ε, Επιτροπής Εποπτείας, αλλά σε συστάσεις του Όλαφ προς τα κρατημέλη. Αυτό είδα πως ε, ανησύχησε αρκετούς από εσάς. Όλαφ λοιπόν διατυπώνει κάποιες συστάσεις και τα κρατημέλη λένε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να πάμε στο δικαστήριο. Αυτό για μας αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να βελτιώσουμε. Ε, να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Όλαφ, διότι ο Όλαφ δίνει τους φακέλους με τα στοιχεία στα κράτη-μέλη και θέλει αυτά να ληφθούν υπόψη από τις εθνικές αρχές. Αυτό δηλαδή ήθελα να πω. Πέτρη. Ναι, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά θέλω να τονίσω ότι η σύσταση που διατυπώνεται είναι κάτι που πρέπει, πρέπει να γίνει, θέλουμε να το δούμε. Συμφωνώ δηλαδή με αυτό που λέτε. Αλλά, επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Ε, υπάρχει και κάτι άλλο στην παράγραφο 48 και την παράγραφο 49 που είναι ακόμα πιο έντονα διατυπωμένο για το νέο σύστημα υποβολής αναφορών που αναφέρει με αρκετά έντονη γλώσσα. Στην παράγραφο 49 αυτό που λέει ότι η Επιτροπή ανησυχεί έντονα, ανησύχησε έντονα από την απάντηση του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ τα λοιπά Αυτό έτσι μου έκανε εντύπωση. Ναι, όπως είπαμε και στην έκθεσή μας, μας ανησύχησε, μας εξέπληξε αυτή η αντίδραση. Βέβαια, στο μεταξύ υπήρξε μία επικοινωνία και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί μια συμφωνία σύντομα. Είμαστε λοιπόν σχετικά αισιόδοξοι ότι θα πάρουμε απαντήσεις. Ωραία, αυτό ήθελα να μάθω. Είχαμε κάποια προβλήματα με την προστασία των δεδομένων, τα οποία χρειάζεται να επιληθούν και πρέπει να τηρήσουμε ε, τα όσα προβλέπει ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Δεν μπορούμε να ε, πούμε ότι λύσαμε τελείως το πρόβλημα, όμως ε, είμαστε καθοδόν, νομίζω σε καλό δρόμο. Ελπίζω μέχρι το 2020 λοιπόν να είμαστε σε θέση να δώσουμε μια θετική απάντηση, μια λύση σε αυτό. Και εμείς το ελπίζουμε. Κύριε Γενική Διευθυντή, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να σχολιάσω τα όσα υπόθηκαν. Καταρχάς να συμφωνήσω με τον κύριο Μάλντερ. Οι συζητήσεις ήταν ανοιχτές. Συχνές. Συζητήσαμε ευθέως το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και πώς ε, πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Στην έκθεση αναφέρεται βέβαια ότι η Επιτροπή ε, εξεπλάγει και εγώ εκπλήσωμαι που το διαβάζω αυτό. Το είπα και στην Επιτροπή ότι θα δώσω όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως προβλέπει ο νόμος. Υπάρχει βέβαια ακόμα μία εκκρεμότητα αυτή της προστασίας των δεδομένων. Υπάρχει ο επόπτης προστασίας δεδομένων, ο οποίος έχει στείλει μία επιστολή για το πώς πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα. Κατά τα άλλα, νομίζω πω ε, αναφέρθηκα σε όλα πω η Επιτροπή Εποπτεία έχει πλήρη πρόσβαση στι υποθέσει, μπορεί να ε, πάρει ό,τι στοιχείο θέλει, όμω Ακόμα και μετά από τη συζήτηση που είχαμε, ζήτησα από τους αρμόδιους μία απάντηση, μία εξήγηση για το τι εννοούν. Οπότε ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα σύντομα. Και εμείς χαιρόμαστε ε, για αυτή τη λύση που φαίνεται στον ορίζοντα. Γιάννη. Προτού φύγετε από την αίθουσα, μάλλον όσο λείπατε. Είπα ότι είχα πολύ καλή συνεργασία με την ε, προηγούμενη πρόεδρο της Επιτροπής σας, την ε, κυρία Γκρέσλε, και ελπίζω υπό τη δική σας προεδρία να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία. Ε, είπα λοιπόν ότι είμαι αισιόδοξο, ότι όσο μάλλον είμαι αισιόδοξο για αρκετέ υποθέσει, είμαι αισιόδοξο και για το μέλλον τη συνεργασία μα. Ε, Γιάν, με συγχωρείς που έπρεπε να καταλήψω την αίθουσα, λέει η συνάδελφος Γκαρθία μου νιώθετε ικανότατη στα καθήκοντα της ε, Προέδρου και εγώ χαίρομαι για την συνεργασία που θα έχουμε. Η κυρία Γκρέσλε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής και συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά μαζί σας προτού αλλάξει ηγεσία Όλα. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσω αυτήν την παράδοση της ε, καλής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόταση αυτή, την οποία δέχομαι ευχαρίστω. Νομίζω πως όλοι τώρα έχετε ξαντληθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον Γενικό Διευθυντή του Όλαφ, όλο και ε, το επιτελείο τους, αλλά και τον αγαπητό Γιάννα Μούλντερ, Σας εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια. Τώρα, πρωτού τελειώσουμε, πριν φύγετε όλοι, να σας ενημερώσω για την επόμενη συνάντηση των συντονιστών 12 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Σας ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών 12 Σεπτεμβρίου από τις 9 τις 10 το πρωί. Σας παρακαλώ να είστε όλοι εκεί. Και αύριο το πρωί, μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού, θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση για την ε, χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Euronews. Σας εύχομαι λοιπόν καλό απόγευμα και καλή ξεκούραση.